We have to elect the new Bureau Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εγώ θα προεδρεύσω σε προσωρινή βάση, γιατί οι κανόνες προβλέπουν ότι ο προηγούμενος πρόεδρος ή η προηγούμενη πρόεδρος θα προεδρεύσει το πρώτο αυτό κομμάτι. Συνεπώς, η συνεδρίασή μας ξεκινάει επίσημα. Δεύτερον, όπως ε, σας είπα ήδη, το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας σήμερα είναι οι εκλογές. Πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο ή την πρόεδρο και μετά τέσσερις αντιπροέδρους. Έναν προς ένα ο κάθε ένας από τους αντιπροέδρους, άνδρες ή γυναίκες, θα εκλεγεί ξεχωριστά. Ε, να έχετε τις κάρτες μαζί σας, μήπως χρειαστούμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Και εφόσον όλα είναι ξεκάθαρα, θα ξεκινήσουμε με τη θέση του Προέδρου. Η απαρτία είναι δεδομένη άνω του 50% των μελών είναι παρόντες. Ακούστηκε κάποιο σχόλιο εκτός μικροφώνου. Και τώρα θα ζητήσω από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να ονομάσουν τον υποψήφιό τους για την Προεδρία της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Έχουμε, λέει ο κύριος Βαν Μίτεμπεργκ, η κυρία Μιχάλοβα που ήδη προεδρεύει ε, και επιθυμεί να παραμείνει για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Η υποψηφία μας λοιπόν είναι η κυρία Μιχάλοβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες προτάσεις, οι υπόλοιποι συντονιστές, όχι, σας ευχαριστώ. Λέει η πρόεδρος, η ιδιταίος και μέλουσα πρόεδρος. Να μου επιτρέψετε όμως να πω εδώ ότι εδώ και δυόμιση χρόνια με υποστηρίξατε χωρίς να με γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε. Την αισθάνθηκα την υποστήριξή σας τα τελευταία δυόμιση χρόνια από όλους τους συναδέλφους και όλες τις πολιτικές ομάδες. Η τιμή ήταν μεγάλη, η χαρά ήταν μεγάλη και θα συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, να συνεχίσω την προσπάθεια σεβόμενη τις απόψεις σας, τις πολιτικές σας θέσεις και την εμπειρογνωμοσύνη σας. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη σε όλους. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρετε πόσο ε, σύντομη ήταν η διαδικασία του Προέδρου. Έχουμε τώρα τις διαδικασίες εκλογής των Αντιπροέδρων. Θα ξεκινήσουμε με την εκλογή του πρώτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ρέτζη. Οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων θα πρέπει παρακαλώ να μας δώσουν τα ονόματα των υποψηφίων. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Καταρχάς συγχαρητήρια λέει ο κύριος Βανίστελ Είχαμε καλή συνεργασία και θα συνεχίσουμε. Τώρα, για τον υποψήφιο. Είναι πίσω μου. Ο κύριος Ζέλα, ο Γερμανός συνάδελφος, ε, έχει οριστεί από την ομάδα μου ως υποψήφιος πρώτος αντιπρόεδρος. Είστε βέβαιος κύριε Βανίστελ Ρόι. Για κοιτάξτε πάλι. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, θα προλάβουμε, θα γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω. Ε, τώρα θα ασχοληθούμε με τον πρώτο αντιπρόεδρο, κυρία Μίσελ. Καταρχήν, ε, θερμά συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε και ελπίζουμε σε μια περαιτέρω καλή συνεργασία. Εμείς από την ΚΟΕΒ προτείνουμε τον κύριο Γιούνο Σομαζή ως ε, υποψήφιο αντιπρόεδρο, δεύτερο αντιπρόεδρο. Λυπάμαι, ως πρώτο αντιπρόεδρο. Okay. Finally we... Ωραία λοιπόν, τελικά έχουμε τις υποψηφιότητες για τον πρώτο αντιπρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, άλλες προτάσεις για τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών. Ε, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, συγγνώμη. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Συγχαρητήρια, κύριε Μαζέ. Παρακαλώ, ελάτε. Και τώρα θα έρθουμε και μπορούμε να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο στην εκλογή του Δευτέρου Αντιπρόεδρου, κύριε Βανίστο ο Γιώχαμ Ζέλαρ από τη Γερμανία έχει ήδη προταθεί. Υπάρχουν άλλες ε, προτάσεις, όχι. Ωραία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κύριε Τσέλερ. Παρακαλώ ελάτε κι εσείς. Και τώρα θα περάσουμε στην εκλογή του τρίτου αντιπρόεδρου. Υπάρχουν προτάσεις για τον τρίτο αντιπρόεδρο, κύριε Βαν Νιστερόι. Ο Πασκάλ Αντεμό, ο Βέλγος συνάδελφος. Θα ήθελα να τον προτείνω. Υπάρχουν άλλες προτάσεις για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Όχι. Συγχαρητήρια, κυρία Αντεμό. Παρακαλώ, περάστε και εσείς στο Προεδρείο της Επιτροπής μας και τώρα θα περάσουμε στην εκλογή του τετάρτου Αντιπροέδρου. Κυρία Γκρέν. Ναι, βεβαίως ε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ εσάς και τους τρεις ε, πρώτους Αντιπροέδρους. Ε, η δική μας πολιτική ομάδα έχει τη μεγάλη τιμή και χαρά να προτείνει τον Ανδρέα Κοσιλίνο και νομίζω ότι πραγματικά μπορεί, ταιριάζει απόλυτα σε όλους εσάς στο Προεδρείο. Υπάρχουν άλλες προτάσεις για τη θέση του τάρτου αντιπρόεδρου. Όχι. Κύριε Κατσουλίνο, θερμά συγχαρητήρια και σε εσά. Παρακαλώ, ελάτε στη θέση σας στο Προεδρείο της Επιτροπής κρύβανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Για τη δική μου πολιτική ομάδα εκ μέρου τη δική πολιτική ομάδα θα ήθελα να πω ότι συγχαίρω του αντιπροέδρου, βεβαίω του στηρίζουμε όλου, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την, ε, με την ε, αναλογία των φίλων. Ε, συνολικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο η εικόνα είναι αρνητική όσον αφορά την ισορροπία των δύο φύλων. Κατ' ουσία μέσω του κανονισμού ε, είμαστε υποχρεωμένοι από το 2014 να την τηρήσουμε. Ε, και θα ήθελα να πω ότι τελικά δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα ήταν αναγκαίο και στη δική μας επιτροπή, όπως και στις άλλες επιτροπές, να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, μια πρώτα σχέση με την ισορροπία των δύο φίλων και να τη στηρίξουμε μελλοντικά. Ε, πέρα από αυτό, ε, βεβαίως ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής μας ότι η προαλή σας εκπροσωπεί την Επιτροπή μας, την υποομάδα για την ισορροπία των φύλων και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, παρατήρησή σας. Στην προσεχή μας συνεδρίαση των συντονιστών θα υπάρξει δυνατότητα να συζητηθεί ε, το σχέδιο ενός μελλοντικού προγράμματος για την εξασφάλιση της ισορροπίας των φύλων μελλοντικά. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ε, όχι. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη της τακτικής μας συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση των πρακτικών. Υπάρχουν καθόλου παρατηρήσεις? Όχι. Άρα λοιπόν εγκρίνουμε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίασή μας και θα ξεκινήσουμε την έγκριση των πρακτικών συνεδρίασης τον 3 ε, Οκτωβρίου 2016, 8 Νοεμβρίου 2016, 9 και 10 Νοεμβρίου 2016 και 29 Νοεμβρίου 2016. Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά ε, online. υπάρχουν και στάσει των συντονιστών για την συνεδρίαση της 29 Νοεμβρίου και της 11 Νοεμβρίου, τα οποία θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μέσω email. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια εδώ, θα σας πρότεινα, εκτό αν υπάρχουν κάποιες ε, ενστάσεις, ε, να προχωρήσουμε στην έγκριση των ε, πρακτικών των συντονιστών και των συνεδριάσεων αυτών. Επόμενο σημείο είναι η ανακοινώση της Προέδρου. Την πιο σημαντική ανακοίνωσή μου την έχω ήδη κάνει. Είπα πόσο χαρούμενη είμαι ε, που θα συνεργαστώ μαζί σας και στη συνέχεια, αλλά έχω και μια άλλη ανακοίνωση που σχετίζεται με τα διάφορα. Όπως σας ενημέρωσα στις 29 Νοεμβρίου η Επιτροπή μας ε, ενέκρινε την Επιτροπή του κυρίου Ισερβάν Ντερόι και της κυρίας Βαν Κρέλ για, την, ε, για διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις με μια πλατιά πλειοψηφία και θα ξεκινήσουν κάποιες διαπραγματεύσεις διοργανικές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και εγκρίνουμε, θα πρέπει να εγκριθεί εντολή για την ομάδα διαπραγμάτευση εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πρώτη συνάντηση έγινε στις ε, 11 Ιανουαρίου του 2017 οι διαπραγματεύσει έγιναν με ένα πνεύμα καλή συνεργασία εν ώψη της ε, μιας ε, ε, ταχείας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και την έγκριση του κανονισμού. Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης κάποια κοινά σημεία και διαφοροποίησει εντοπίστηκαν και τέθηκαν τα βασικά ερωτήματα σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Μετά την πρόταση της Γραμματείας της Επιτροπής Περιφυγής Ανάπτυξης, η συζήτηση ε, επικεντρώθηκε γύρω από βασικά θέματα της εντολής του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις δραστηριότητε, της ομάδας, των προγράμματος εργασίας και της εφαρμογής καθώς και της, ε, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ε, στο τέλος αυτής της πρώτης συνεδρίασης οι συμμετέχοντες ε, συμφώνησαν πολλά θέματα να διαβιβαστούν, ε, να μεταφερθούν στις τεχνικές συνεδριάσεις τους ώστε να διευκολυνθεί η προσοχή μας συνεδρίαση. Η επόμενη τριμερή συνάντηση έχει προγραμματιθεί για τις 25 και 31 Ιανουαρίου του 2017 και θα σας αναφέρουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίας, προσοχή μας συνεδρίαση. Αυτά για, την, για το πρόγραμμα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχετε καθόλου σχόλια. Όχι. Και τώρα θα περάσουμε στην εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης που προετοίμασε ο συγητής μας κύριος Μπρέσελ για την ε, παράταση της εντολής ε, για τις στρατηγικές επενδύσεις Έχετε το λόγο κυρία Μπρέσαλ. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για την εκλογή σας λέει κυρία Μπρέσο. Θα συνεχίσω Ιταλικά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα την προσπάθεια την οποία έκανα για την γνωμοδέτησή μας ε, για την παράταση λειτουργίας του ΕΦΣΥ και τις τροποποίησης του κανονισμού της σχετικές με την Επιτροπή μας. Περιορίστηκα δηλαδή στα θέματα τα οποία μας αφορούν, γιατί αλλιώς γνωρίζετε ότι οι προτάσεις μας δεν θα γίνουν δεκτές από τις κύριες επιτροπές. Θα είμαι σύντομη και θα σας δώσω την δυνατότητα να μου μεταφέρετε τις δικές σας παρατηρήσεις και συστάσεις. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι το στρατηγικό ταμείο επηρέασε με συγκεκριμένο και θετικό τρόπο τις οικονομίες μας. Νομίζω ότι ήταν μια πρώτη και σημαντική εξ αυτού πρωτοβουλία είναι μια νέα εποχή ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδέχεται ότι πέρα των ιδιωτικών επενδύσεων μια δημόσια παρέμβαση μέσω χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό λοιπόν είναι ουσιώδες να συνεχιστεί το Ταμείο αυτό και στο άμεσο μέλλον όπως ακριβώς προτείνεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι πεπισμένη που απαιτείται μια ανάκαμψη του Ταμείου αυτού με περισσότερους πόρους και με ρυθμίσεις επιμέρους όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα. Είναι σαφές βέβαια ότι δεν μπορούμε εμείς να σκεφτούμε το εύση ε, σαν κάτι το οποίο μονίμως θα αφαιρεί χρηματοδοτήσεις από άλλα προγράμματα που είναι και αυτά σημαντικά για πολλούς πολίτες μας και τα οποία λειτουργούν ε, κανονικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ήπειρο. Συνεπώς λοιπόν το θέμα των ιδίων πόρων παραμένει χένον, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα ε, μέσα στα δεδομένα όρια που θα πρέπει να αυξηθούν για να αυξηθούν και οι επενδύσεις. Πάντως έτσι όπως έχουν τα πράγματα εγώ προσπάθησα με χειρουργικό τρόπο να δράσω επεμβαίνοντας όπου μόνον αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε το κείμενό μας να μεταφέρει το συγκεκριμένο μήνυμα της δουλειάς την οποία κάνουμε όπως και οι άλλες επιτροπές. Ξέρετε ότι πρόκειται για έναν κανονισμό όπως σας είπα λοιπόν, κατέθεσα και τροπολογίες μέσω των οποίων αφού τις ψηφίσουμε θα προσπαθήσουμε να περάσουν από τις κύριες επί της ουσίας δηλαδή κοινοβουλευτικές επιτροπές. Καταρχάς, εγώ υπογράμμισα την πάρα πολύ μεγάλη σημασία την οποία έχει μια βελτιωμένη συνέργεια ανάμεσα στο ΕΦΣΙ από τη μία και τα τα ταμεία από την άλλη. Διαφορετικά ταμεία, διαφορετικοί στόχοι, τα μεν για τις πολιτικές μας πιο αποτελεσματικές, το άλλο για περισσότερες επενδύσεις. Αλλά είναι απαραίτητο να συντονιστούν έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους τους κοινού αηφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής, εδαφικής και οικονομικής συνοχής. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δοθούν περισσότερες εγγυήσεις για την συμπληρωματικότητα των δύο αυτών μέσων, και γυρνιάζοντας το περιεχόμενο των λογιστικών κανονισμών, διότι ακριβώς οι λογιστικές ρυθμίσεις για κάθε ταμείο λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και καθιστούν τη συγκρισιμότητα δύσκολη και θα πρέπει μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων να καταλήξουμε σε μια καλύτερη γεωγραφική κάλυψη του εδάφους της Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ορίσουμε ποσοστώσεις αναχώρα. Μιλάμε και για ιδιωτικές επενδύσεις και για ποιοτικέ επενδύσεις και θα ήταν λάθος κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερα μέσα στις αρμόδιες αρχές ενισχύοντας τις δυνατότητες επιλογής, ενισχύοντας την τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη, έτσι ώστε διατηρώντας το Ταμείο ανοιχτό και ποιοτικό, να μπορέσουν οι επιμέρους χώρες να πάρουν μεγαλύτερο μέρος από ό,τι στο παρελθόν. Ένα από τα σημαντικά σημεία του ΕΦΣΙ θα είναι η εγγύηση της προσθετικότητας των προγραμμάτων που υποστηρίζονται. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν ενισχύοντας τον ρόλο των συμβούλων επένδυσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένες μικρές χώρες μπορεί να έχουν και αυτές μια περιφερειακή πλατφόρμα συμβούλων. Οι πλατφόρμες αυτές ε, πρέπει να είναι χρήσιμες γιατί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα τις ανάγκες των συγκεκριμένων ε, περιοχών και μπορούν να είναι κοντά στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό δούλεψε ακριτά καλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι τόσο για τις υπόλοιπες. Τα κράτη λοιπόν είναι παρόντα στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΦΣΥ και με τα ποσοστά τα προκαθορισμένα εκ των προτέρων. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν καλύτερα τις υπεύθυνε αρχές και τους διαχειριστές του Ταμείου στον τομέα των χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία θα εγγυηθούν την πλήρη επιτυχία της πρωτοβουλίας ΕΦΣΗ. Πολλές φορές η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και για τα διαφορετικά ταμεία μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να συνδυαθούν οι δύο παρεμβάσεις. Σαν παράδειγμα ακούσαμε τον πρόεδρο ε, του, τον πρόεδρο των περιφερειακών ε, θαλάσσιων περιοχών, παραθαλάσσιων περιοχών, ο οποίος είπε ότι συνδυάζοντας ε, τα διαφορετικά ταμεία και τα εύση σε μεγάλα προγράμματα υποδομών πετυχαίνει κανείς καλό αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητο λοιπόν τα μέσα αυτά να μπορέσουν να καταφέρουν να συγκλίνουν μέσω των κανονισμών τους και όχι να αποκλίνουν. Λοιπόν αυτά είναι χοντρικά αυτά που θα ήθελα να σας πω. Έχετε ένα πιο συγκεκριμένο κείμενο στην διάθεσή σας και έχετε επίσης και τις τροπολογίες τις οποίες σας προτείνω. Είμαι αν θέλετε στη διάθεσή σας για να σχολιάσω τις παρατηρήσεις σας και να προσαρμόσω το κείμενο επί τη βάση της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τους της συζήτητας. Ο κύριος Ντάτ. Είναι πρώτος συζήτης. Σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν είναι καινή τυπικότητα αυτό. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Πρόεδρο και τους αντιπρόεδρους για την επανεκλογή τους. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας εύχομαι επικοδομητική εργασία για τα επόμενα δύο και δυόμιση χρόνια. Και τώρα να κοιτάξουμε το σχέδιο έκτασης της κυρίας Μπρέσσαου. Επιτρέψτε μου να διατρέξω τις ιδέες μία προς μία. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τις απόψεις του ΕΛΚ και θα πρέπει καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι το ΕΦΣΥ ένα έτος μετά την θέση του σε εφαρμογή βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει πρόταση για να παραταθεί η διάρκεια ισχύω ε, του Ταμείου, να αυξηθούν οι πόροι και να ενισχυθεί η υποστήριξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μας σημαίνει ότι κανείς δεν έχει αξιολογήσει πραγματικά το πώ έχει λειτουργήσει το ΕΦΣΥ το πρώτο έτος. Υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει την πρόταση αυτή χωρί να έχει κάνει ει βάθο αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μιλούν λοιπόν για την παράταση της ισχύω του, για την αύξηση των πόρων, την διεύρυνση των ε, στόχων και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή όπου κανείς δεν έχει, επαναλαμβάνω, κάνει ενδελεχή αξιολόγηση του Ταμείου. Ούτε η Επιτροπή, ούτε το Κοινοβούλιο ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημείο που ήθελα να αναφέρω. Κάτι άλλο. Τώρα, κατά δεύτερον, το είπε και η κυρία Μπρέσο στην εισαγωγή τη. Έχοντα εξετάσει το σχέδιο έκθεση, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, πολλέ ε, επικοδομητικέ προτάσει, τι οποίε και υποστηρίζουμε. Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα τα οποία αναφέρει η κυρία Μπρέσο είναι το εξή. Το ΕΨΙ και το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει την ε, αξιοποίηση του Ταμείου δεν έχει γεωγραφική κατανομή. Και φυσικά όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ διευθυντικών ταμείων και εύση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ξέρουμε πως ε, διαφέρουν στον τρόπο λειτουργίας τους και ασφαλώς δεν ε, διατηνόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρχουν φάκελοι για το κάθε κρατός μέλος στα πλαίσια του Εύση. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ταμείου. Έως τώρα, από γεωγραφικής άποψης δεν υπάρχει σωστή κατανομή. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τα project και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν το 2004 για να αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε επίπεδο των κρατημέλη αυτά σε 90% σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εγγύησεις που δίνει το ΕΦΣΥ. 90% δηλαδή πηγαίνει στα κρατημέλη που είχαν προσχωρήσει πριν από το 2004 ή άλλες χώρες, αυτές που μπήκαν μετά το 2004 δηλαδή, αξιοποιούν μόνο το 10% των πόρων αυτών. Περίπου τέλο πάντων, συγχωρέστε με, δεν είμαι 100% ακριβής. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Αν ε, δούμε ποια είναι η χρηματοδότηση κατά κεφαλή, είναι 20.000 ευρώ ανά άτομο και 7.000 και 7 ευρώ στις δύο αυτές ε, κατηγορίες που σας είπα, δηλαδή για κάθε πολίτη από τα παλιά κρατημέλη 20.000 ευρώ και 7 ευρώ κατά κεφαλή για τους πολίτες των νέων κρατών μελών. Αυτό το πρόβλημα θεωρώ ότι αποτελεί και την αιτία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Χαιρόμαστε που η κυρία Μπρέσαου επιχειρεί να διορθώσει το πρόβλημα αυτό και θα θέλαμε από πλευρά του ΕΛΚ να καταθέσουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. ανέφερα πώς θα βελτιωθεί η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει ήδη αυξηθεί η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήταν απαιτικό αυτό το αποτέλεσμα και το ΕΦΣΙ πραγματικά σημείωσε επιτυχίες ω προ την άποψη αυτή. Να μην σα κουράσω με στατιστικά στοιχεία. Όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. όπου δεν αποτελούν ραχοκοκαλιά της οικονομίας ή μικρομεσαίες. Παντού ισχύει αυτό. Χρειάζονται λοιπόν κίνητρα, χρειάζεται υποστήριξη των εταιρείων αυτών. Γιατί αυτές είναι που τονώνουν το ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο στοιχείο τώρα, κάτι που επίσης ανέφερε η κυρία Μπρέσαου, η σχέση μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και ταμείου στρατηγικών επενδύσεων εύση. Ίσως αυτό. Καλό θα κάναμε να το υπογραμμίζαμε λίγο παραπάνω. Η εναρμόνιση, ο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και του ΕΦΣΥ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλός. Ωστόσο, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο εν μέρη προέρχεται από έλλειψη συνεργειών και εν μέρη λόγω των διαφορών σε ό,τι αφορά των προσεγγίσεων για τη χρήση των δύο ταμείων. Δεν λέω είναι αντίθετα τα ταμεία και οι προσεγγίσει τους, αλλά σε κάποιε περιπτώσει ο κόσμο θεωρεί ότι είναι εναλλακτικά αυτά τα ταμεία, ή το ένα ή το άλλο δηλαδή. Ότι είναι διαζευτική έτσι η χρήση τους. Θα πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό όταν τροποποιήσουμε τον κανονισμό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η αύξηση και των πόρων και της διάρκειας ε, του Ταμείου Επενδύσεων, του ΕΦΣΥ, δεν θα σημαίνει ούτε τώρα, ούτε μετά το 2020, ότι αποτελεί αυτό εναλλακτικό ταμείο ω προς τα ταμεία. Και εμείς από την ε, Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η πολιτική συνοχής κατοχυρώνεται στη συνθήκη και θα συνεχιστεί μετά το 2020. Αυτή είναι η αφετηρία, του σημείου κίνησή μας, το εύση, είναι κάτι συμπληρωματικό, μια πρόσθετη αξία. Ποτέ όμως δεν πρόκειται να αντικαταστήσει. Αυτά λοιπόν τα σχόλια ως προς ε, τα όσα μας παρουσίασε η κυρία Μπρέσα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και προφανώς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Η κυρία Τόμασιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σα συγχαρώ και εγώ για την επανεκλογή σα. και στους υπόλοιπους, ε, στους αντιπρόεδρους να πω συγχαρητήρια. Να σας πω ότι αισθάνομαι ότι είμαι σε οικογενειακό περιβάλλον εδώ στην Επιτροπή μας ε, και υποστηρίζω την εισηγήτρια, την κυρία Μπρέσα. Η γνωμοδότηση λοιπόν της Επιτροπή μας για την παράταση του ΕΦΣΥ θεωρώ ότι σκοπό έχει να εξασφαλίσει την ε, στον συντονισμό μεταξύ των ταμείων και της συμπληρωματικότητα. Η υποστήριξη λοιπόν των διαφόρων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να ε, προκαλεί διπλή και τριπλή δουλειά. Όχι, θα πρέπει από κάθε ταμείο να υπάρχει μια πρόσθετη αξία. Και θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με τις περιφερειακές και εθνικές τράπεζες ανάπτυξης και επενδύσεων η συμπληρωματικότητα λοιπόν μεταξύ του ΕΦΣΙ και των ιερωτικών ταμείων θα μπορούσε να δώσει έναυσμα και στις επενδύσεις. Και αυτό λοιπόν περιλαμβάνεται και στο σημείο 1. Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσει τη Τράπεζα Επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών. Θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται τεχνική υποστήριξη για τη διάρθρωση α, της α, ε, χρηματικής και θα πρέπει να εστιαστούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις ε, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και κυρίως να λοιπόν υπόψη τα κρατημέλη όπου η αγορά είναι λιγότερο αναπτυγμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α, ενημερώνεται για όλες τις νομοθετικές προτάσεις και έτσι υπάρχει σωστή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι η επόμενη σκιώδη εισηγήτρια. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω βουλγάρικα, αν μου το επιτρέπετε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσαου за изготвеното становище по предложения регламент. ευχαριστώ λοιπόν κυρία Μπρέσα για την γνωμοδότηση αυτή. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά την παράταση των δραστηριοτήτων του ΕΦΣΥ όπως και την αύξηση των οικονομικών πόρων. Αναφέρεται επίσης και σε κάποιες τροποποιήσεις της δραστηριότητας του Ταμείου. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας μπορούμε να μιλήσουμε για δυνατότητες βελτιώσεων. Μετά από την σύντομη παρουσία του Ταμείου, κάποιες παρατηρήσεις μπορεί να γίνουν, ιδιαίτερα δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών και πιέσεων Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να προσελκύουμε κεφάλαια σε προγράμματα, κάτι το οποίο θα επιτρέψει τη δημιουργία εθνικών πόλων που θα, χρηματοδοτούνται από τα παλαιότερα ταμεία και από το νέο ταμείο. Και γι' αυτό εδώ υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Μπρέσο για καλύτερες μορφές συντονισμού και περισσότερο συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα ταμεία. Αυτός είναι ο δρόμος για την μεγέθυνση των επενδύσεων και την κάλυψη των αναγκών. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το Ταμείο αυτό να λειτουργήσει και για διαμεθοριακά προγράμματα διότι τα διαμεθοριακά προγράμματα είναι σαφώς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας από τα αυστηρά εθνικά. Έχει σημασία λοιπόν να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σύμβουλων και να ενισχύσουμε και την δημιουργία του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε το Ταμείο αυτό να λειτουργήσει σωστά στο μέλλον. θα μπορέσουμε μέσω των εθνικών αυτών πόλων να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες στρατηγικής σημασίας και γι' αυτό θα υποστηρίξω και τις τροποποιήσεις, τροπολογίες καλύτερα, τις οποίες προτείνει η κυρία Μπρέσο για τη λειτουργία του Κέντρου Διαβούλευσης. Να υποστηρίξω λοιπόν την γνωμοδότηση της κυρίας Μπρέσο γιατί πράγματι στοχεύει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας, της δράσης του Ταμείου και στον καλύτερο συνδυασμό του Ταμείου αυτού με τα διαφθρωτικά ταμεία. Εδώ να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο, να εμπλέκονται περισσότερο στη λειτουργία του Ταμείου και να εμπλέκονται επίσης και στην λειτουργία και τις δραστηριότητες των εθνικών πόλων. <clears throat> να πω παράλληλα ότι η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΦΣΥ <clears throat> θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και τις πιθανές αλλαγές σε αυτό δηλαδή σε πολιετή βάση και αυτό ισχύει κυρίως για την περίοδο μετά το 2020. Η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και γι' αυτό υποστηρίζω για μια ακόμη φορά την πρόταση Μπρέσο. Μίχελ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να κρύψω ότι από τη δική μου πλευρά, πολιτική ομάδα, έχουμε κάποιες αμφιβολίες ε, σχέση με το κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη χρονική στιγμή ήδη ένα χρόνο μετά τη θέση ισχύ της πρωτοβουλίας για μια παράταση, να μιλούμε για μια ε, ε, παράταση της, ε, της λειτουργίας του ΕΦΣΥ. σε μια γνωμοδότησή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας είπε ότι δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ότι η προταθήσα αύξηση των κονδυλίων είναι δικαιολογημένη και ενδεχομένως ε, δεν μπορεί να υπάρξει και μια μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων και συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε εντιμότητα όσον αφορά την ε, αξιολόγηση λειτουργίας του ΕΦΣΥ και στη Γερμανία είχαμε ανταλλαγή απόψεων με πολλά ομόσπονδα κρατήδια, τα οποία όλα θεωρούν ότι το ΕΦΣΥ το οποίο είναι προσανατολισμένο σε μεγάλα, μεγάλες εμβέλειες προγράμματα, ε, δεν ε, καλύπτει τις ε, περιφερειακές ανάγκες και δεν είναι αποτελεσματικό όσον αφορά τη δημιουργία συνεργειών. Γιατί τα μεγάλα προγράμματα και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε έντιμοι και να μπορούμε έντιμα ειλικρινά να το αξιολογήσουμε τα μεγάλα προγράμματα στις περιφέρειες που πραγματικά έχουν ανάγκη δεν φτάνουν και τα κριτήρια πρόθεσης έχουν οριστεί ε, πολύ ε, χαλαρά και δεν, ε, πολύ αόριστα και δεν θεωρούμε και θεωρούμε ότι πραγματικά είναι κρίσιμο το ζήτημα διασύνδεσης με το Διορθωτικό Ταμείο, γιατί κατά την άποψή μας εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, η βασική ιδέα των δημόσιων υπηρεσιών και των ε, δημόσιων υποδομών τελικά να αντιστραφεί και ως εκ τούτου δεν μπορώ να μοιραστώ αυτή την ε, πολύ, ε, αυτό το πολύ αισιόδοξο πνεύμα που κυριαρχεί εδώ. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει η αξιολόγηση και όχι να εγκρίνουμε την παράταση ε, ξεκινώντας από τα πράγματα όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία συνάδελφε, ε, εκτιμώ πάρα πολύ την εργασία σας ως συγγήτριας, την εκτιμώ εξαιρετικά, αλλά και εμείς συριζόμαστε την ε, κριτική της ε, σε συναδέλφου. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να μοιραστούμε την ε, βασικά θετική εκτίμηση του ΕΦΣΙ. Γιατί για μας ήδη όσον αφορά τη λογική της οικοδόμησης του ΕΦΣΙ βλέπουμε ότι εδώ υπονομεύονται οι στόχοι της πολιτικής συνοχής. Και δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραταθεί η λειτουργία του. Ιδιαίτερα η μη διασύνδεση μεταξύ ποιοτικών στόχων, μόνο 4% των κονδυλίων ε, πάνε σε προγράμματα υποδομών ε, και σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Τα περισσότερα προγράμματα ε, αντιβαίνουν μάλιστα στους στόχους της Ευρώπης 2020. Και αυτό μας έχει υποσχεθεί στο παρελθόν ο αντιπρόεδρος κ. Κατάινεν. Και είδαμε ότι, επίσης ότι η αύξηση της απασχόλησης επιτυχάνεται μόνο εφόσον γίνονται επενδύσει σε περιοχέ όπου υπάρχει μεγάλη φτώχεια και ανεργία. Και δεν βλέπω αυτή η σκέψη να έχει ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προγραμμάτων. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ για τα επενδυτικά ταμεία τελικά να αφαιρούν πραγματικά χωρίς όρια, περιόριστα κάποια κονδύλια από τα διευθυντικά τομεία. Ε, και για μας αυτό σηματοδοτεί το τέλος της διευθυντικής πολιτικής, το τέλος ε, της βάσης μιας κοινωνικής οικονομίας και μιας κοινωνικής συνοχής που είναι ο πρώτος το στόχος της πολιτικής συνοχής και σηματοδοτεί επίσης το τέλος των ε, ολοκληρωμένων ε, προγραμμάτων ε, συνοχής και της συμπεριλήψης όλων των διαφορετικών φορέων. Και θα ήθελα να τονίσω και ένα σημείο λέγοντας ότι αξιολογούμε θετικά το βήμα ότι 20% των κονδυλίων του ΕΦΣΥ που πάνε σε επενδύσει και καινοτομίε θα συνδεθούν με περιβαλλοντικούς στόχους. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και θα είμαστε μάλιστα υπέρ ενός 50% αντί για το 40% που προβλέπετε εδώ αλλά αυτό θα αφορούσε και μία, θα σε και μία αλλαγή του ΕΦΣΗ. Τώρα, σε τροπολογίες θα ζητήσουμε μία αυξημένη διαφάνεια. Στο μέτρο που εδώ εγκεκριμένα προγράμματα τα οποία έχουν αρτηθεί στην ισοσελίδα ε, της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων και μάλιστα άμεσα μετά την έγκριση των προγραμμάτων βάσει των προτάσεων της Επιτροπής εδώ θα υπάρχει τελικά μία μείωση της διαφάνειας γιατί τα προγράμματα θα δημοσιοποιούνται μόνο μετά την υπογραφή τους. Αλλά όπως όλοι ξέρετε η υπογραφή μπορεί να παραταθεί για πολλούς μήνες, να καθυστερήσει υπερβολικά. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ μια μείωση διαφάνεια όσον αφορά την δημοσιοποίηση των λόγω προγραμμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία με την κυρία Πρεσό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ms. Demato. The floor is yours. Σας ευχαριστώ, κύριε Δεμάτο. Έχετε λόγο. Η κυρία Δεμάτο. Να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ καλή δουλειά στην Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους. Το κίνημα των πέντε αστέρων θα συνεισφέρει, συγγνώμη για την, παρουσία, την απουσία μου προηγουμένως, αλλά ήμουνα στην Επιτροπή Αναφορών, όπου έπρεπε να δούμε να εκλέγεται Ε, ένας εκπρόσωπος των πέντε αστέρων, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό και δεν έγινε σεβαστή η μέθοδος Hont. Ακυρώθηκε η εφαρμογή της μεθόδου Hont. εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια πριν δύο χρόνια είχαμε το άλλο άλοθη ότι δεν μας γνωρίζατε, αλλά τα δυόμιση χρόνια νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές των πέντε αστέρων απέδειξαν ότι είναι συστηματικά προπαρασκευασμένοι και ικανοί να εκπροσωπήσουν τους συμπολίτε τους στο Κοινοβούλιο. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν γιατί σας κάνω να χάσετε το χρόνο σας, αλλά όφιλα να σας το πω αυτό. Να πω ότι η πρόταση για το ΕΦΣΥ προβλέπει ουσιαστικά τη διόρθωση των δύο κανονισμών. Με το άλοφι της συνέργειας και της προσθετικότητας με τις πολιτικές συνοχής το ΕΦΣΥ φτώχινε άλλες δράσεις ε, προϋπάρχουσες όπως ε, και το Εράσμους και άλλα. Πολλές φορές ε, το ΕΦΣΥ στάθηκε αδιαφανές χρηματοδότησε ε, θα έλεγα τεράστια προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αηφορία ε, όχι μόνο ωφελεί τους ενδιαμέσους και τις τράπεζες αλλά ε, αποκρύβει τους τρόπους με τους οποίους χρηματοδοτείται το πρόγραμμα αυτό. Η διεύρυνση λοιπόν του Ταμείου μετά από ένα χρόνο λειτουργίας μόνον βασίζεται πάνω σε πάρα πολύ περιορισμένα στοιχεία και δεν θα το στηρίξουμε διότι θα οδηγήσει σε μια υπερβολή της, α, της μόχλευσης έτσι όπως προβλέπεται. Και θα πρέπει η συγγήτρια να ζητήσει μεγαλύτερη ενημέρωση και καλύτερες επιμέρους πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας. Θυμίζω ότι όχι το κίνημα των πέντε αστέρων, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο λέγει, και το διαβάζω κατά λέξη, ότι οι αυξήσει ε, του, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της ε, σύνδεσης του ΕΦΣΥ με την ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία όμως ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν εμείς ασκούμε κριτική σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έχω τα μέλη, τον κατάλογο των μελών που θέλουν το λόγο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ζέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ζητώ το λόγο τώρα γιατί θέλω να πάω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού που έχουν ε, κάποιες ψηφοφορίες. Σε ό,τι αφορά την παράταση του ΕΕ, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να γίνει μια εντελεχέστερη μελέτη σε πρώτη φάση και εξέταση. Το είπε και η κυρία Μπρέσαου. θα πρέπει να εκφέρουμε μια γνώμη ως Επιτροπή Περιφερειών, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι το ΕΦΣΥ δεν έχει να κάνει με τα διορθωτικά ταμεία. Γιατί ο συνδυασμός των δύο χρηματοδοτικών μέσων είναι πολύ δύσκολο θεωρώ, γιατί τα κράτη και οι, περιφερει... και... οι αποφασίζουν για τα διορθωτικά ταμεία, ενώ το ΕΦΣΥ αποφασίζει μόνο η Τράπεζα Επενδύσεων. Και αυτό αποτελεί μια θεμελιώδη διαφορά. Επόμενο θέμα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Από πού προέρχονται τα χρήματα για την παράταση του Ταμείου. Αν είναι να προέλθουν αυτά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, ξέρετε ότι είναι ήδη παραπεντωμένος. Και δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Βιομηχανίας ή Μεταφορών ε, θα είναι επιτεθειμένοι να δώσουν εδώ πέρα χρήματα από τον ε, Horizon 2020 ε, και από το Connecting Europe. Να τονίσουμε επίσης, ε, θεωρώ ότι το ΕΦΣΥ δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να αποτελέσει ποτέ υποκατάστατο για διαφορετική πολιτική με το 2020 και δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια αντιστάθμιση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη στοχοθέτηση, κοιτώντας τα μεμονωμένα project, ε, Θέλουμε να προωθήσουμε τις αρχικές επενδύσεις. Το μοναδικό έργο που βρήκα στην Ελλάδα είναι 5 εκατομμύρια για μια τεχνολογία ε, μεσογειακής δίαιτας ε, που αφορά τα λίπη, τα κορεσμένα τα οποία προχωρούνται από το κρέας, πώς μπορούν να ε, αντικατασταθούν από πιο υγιή τέτοια λίπη. Τώρα αυτό πώς μπορεί να αποτελεί στρατηγική επένδυση δεν μπορώ να σας πω. Το ΕΦΣΙ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προφανώς ε, έχει συμφέρει με Τράπεζα Επενδύσεων από το ΕΦΣΙ. Εμείς από πλευρά της ε, Επιτροπής μας πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η εφαρμογή του ΕΦΣΙ. Όλα αυτά φυσικά έχουν σωστό σκοπό, αλλά τώρα το τι έχει επιτευχθεί αυτό ως τώρα είναι μάλλον εκκρεμές ακόμα και αβέβαιο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, ο κ. Πότσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σέλερ. Σήμερα πώς μπορούμε να ε, εκτιμήσουμε και να εξελογήσουμε το ΕΦΣΙ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. είναι πάρα πολύ πρόημο. Να πω και το εξή. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως και μετά από πίεση της Επιτροπής μας, κλείνει στην ε, συμπερίληψη της συμπληρωματικότητας των δύο ταμείων. Αλλά, από την άλλη, θεωρώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον η μέθοδος ε, προώθησης της ε, συμπληρωματικότητας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σωστή και σκόπιμη. Από πλευράς της Επιτροπής Περιφερειών που ασχολήθηκε με το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Εγώ θα προσπαθήσω να απλοποιήσω κάπως τη διαμόρφωση της ε, γνωμοδοτήσης ε, με τις ε, τροπολογίες μου. Να ρωτήσω λοιπόν την κυρία Μπρέσα, πώς αποφάσισε να υποστηρίξει αυτή τη συμπληρωματικότητα. Ο επόμενο ομιλητή. ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλου του επανεκλεχθέντες από πλευρά του Προεδρείου και σε πρώτη και καλύτερη γίνηση στην Πρόεδρου. Τώρα θα μιλήσω ρουμάνικα, μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι ότι κάτω από τις ε, συνθήκες οι οποίες διευκρινίζονται καλύτερα θα μπορούσαμε να προτείνουμε την ε, ε, χρονική παράταση του ΕΦΣΥ. Από την άλλη όμως πει να τονίσω ότι ορισμένα στοιχεία του ΕΦΣΥ απαιτείται να επαναξιολογηθούν. Ξεκινώ από την στρατηγική διάσταση του συγκεκριμένου μέσου. Η στρατηγική αυτή διάσταση είναι απαραίτητη. Αν δούμε τον κατάλογο των κατά προτεραιότητα επενδύσεων, δεν βρίσκουμε και πάρα πολλά παραδείγματα, προγράμματα, τα οποία να μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε στρατηγικά. Ο κύριος Τσέλερ είπε πολύ σωστά ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για στρατηγικά προγράμματα όταν μιλάμε για χρηματοδοτήσεις ύψους 5 εκατομμυρίων θα πρέπει μια κάποια μεγαλύτερη αν θέλετε διάσταση στις επενδύσεις να είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να καλυφθεί και το, πρόγραμμα, το πρόβλημα των ανισορροπιών σε γεωγραφικό επίπεδο. Όταν αναλύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το Ταμείο αυτό τον πρώτο χρόνο, διαπιστώνει εύκολα τις πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες οι οποίες πήραν χρήματα και τις υπόλοιπες χώρες. Όπως γνωρίζετε ε, η διαφορά αυτή ε, ξεπερνάει τα 6-7 δις για κάποιες χώρες και τα 10 εκατομμύρια για άλλες χώρες. Ξέρουμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες οι οποίες ε, αποφελούνται από την πολιτική συνοχή και ποιοι είναι οι καθαροί πάροχοι. Ποιες χώρες δηλαδή δίνουν χρήματα και δεν αφαιρούνται σχεδόν καθόλου. Δεν υπάρχει ισορροπία περιφερειακή και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον ταμείο αυτό να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Κάτι άλλο τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάγκη να τονίσουμε το εξή στην παρούσα φάση. Το εύση δεν αποτελεί υποκατάστατο, εναλλακτική, δεν είναι συμπλήρωμα για τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Αν η Επιτροπή μας δεν το τονίσει αυτό και αν δεν αποθαρρύνει και τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία θέλουν να αλλάξουν με ριζοσπαστικό τρόπο την πολιτική συνοχής, αν δεν επαναλάβουμε ξανά και ξανά την ανάγκη να υπάρχει πολιτική συνοχή, δεν ε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να είναι σαφές λοιπόν το τι ισχύει. Τέλος. Είναι ζωτική σημασία να βρούμε και μία απάντηση στις ανάγκες τεχνικής αρρωγής για όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή του Ταμείου. Και γιατί. Γιατί συχνά λέμε ότι υπάρχουν χώρες που μπορούν με άνεση να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο. Μπορούμε όμως στην περίπτωση αυτή να μιλήσουμε για πολιτική συνοχή. Όχι, θα πρέπει να σκεφτούμε και τις ανάγκες των χωρών. Υπάρχει λοιπόν τεράστια ανάγκη για παροχή τεχνικής αρρωγής. Μα άμα συνεχίσουμε τον τρόπο αυτό θα συνεχίσει και θα διαγκωθεί και ο ευρωσκεπτικισμός. Θα θεωρεί ο κόσμος ότι όλα αυτά ωφελούν τους άλλους και όχι τον ίδιο. Και αυτό προφανώς θα αυξήσει την κριτική που ασκούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μια ρεαλιστική προσέγγιση για να επιληθούν όλες αυτές οι διαφορές. Και να συγχαρώ τέλος και την εισηγητρία για το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο είμαι πεπισμένος ότι και με τις ε, χρήσιμες ε, παρεμβάσεις μας και προτάσεις μας θα βελτιωθεί έτη περαιτέρω. Και θα βοηθήσει και το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Ο κ. Μίλτεμπεργκ. Ευχαριστώ καταρχήν. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, καταρχήν για την εκλογή σας. Θα είμαι πολύ σύντομος. Έχω περισσότερο μία ερώτηση παρά μία παρέμβαση. Το ερώτημά μου αφορά την τροπολογία 3 και την τροπολογία 10. Στο αρχικό κείμενο της πρότασης είχα την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εστιάσει στην αποφυγή του να στηρίξει το εύση ε, προγράμματα υποδομών όπου βεβαίω μπορούν να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ως προς την προστατικότητα. Ε, δεν ε, ενέχει να κίνδυνο η τροπολογία 3 και το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία παριθμών 10. Δεν ανοίγεται με αυτό το κουτί της ε, Πανδώρας που χάνεται την εποπτεία αυτών των προγραμμάτων ε, αναφέροντας ε, προγράμματα επενδύσεων σε ε, αυτοκινητοδρόμους σε ολόκληρη την ε, Ευρώπη. Uh, uh, Αλλάζοντα πλήρω το κείμενο και θα αναφερθώ μόνο στην, ε, ε, βιώσιμες, στις βιώσιμες υποδομές βεβαίως κάτι το οποίο είναι βιώσιμο για μια χώρα δεν είναι εξορισμού βιώσιμο και για μια άλλη. Ε, Δεχομένω λοιπόν εγκυμονείται εδώ αυτός ο κίνδυνος μέσω αυτών των ε, τροπολογιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Βαν Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να προσθέσω στη συζήτηση το εξή. Θα πρέπει να τονίσω τα όσα ελέγχθησαν εν σχέση με την ε, κατά πόσο χαλάλη η χρονική στιγμή αυτής της παράτασης. Η Επιτροπή είπε ότι η αξιολόγηση θα γίνει γύρω στο 2018. Εγώ έθεσα ε, κατά επανάληψη αυτό το ερώτημα για την αξιολόγηση ε, δεν πρόκειται για μια σοβαρή αξιολόγηση. Είναι σαν να ε, ρίχνει κανείς ε, έναν ε, πύραυλο και ε, να μην ξέρει καθόλου, να μην παρακολουθεί καθόλου την τροχιά του. Ε, ωστόσο ήταν μια υπόσχεση της Επιτροπής, το οποίο θα προκαλέσει μια χιονοστιβάδα νέων πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποδεκτικά στοιχεία πρόκειται μόνο για την πεποίθηση ότι αν ε, συνεχίσουμε ενδεχομένω με την ίδια τακτική ε, θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Αλλά αν θέλουμε να εμβαθύνουμε, ήταν το θέμα της προστατικότητας το οποίο εισαγάγαμε εδώ, γιατί στην πρώτη πρόταση η προστατικότητα δεν υπήρχε. Ε, πρόκειται για δυτικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Αλλά εμείς προσθέσαμε το στοιχείο της προστατικότητας και νομίζω ότι θα πρέπει να αποδειχθεί. Γιατί εάν ε, επενδυθούν ε, εκατομμύρια ε, σε, ένα, σε μια περιοχή της, σε δίκτυο της Νοτιού Γερμανίας, όπου όμως δεν υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, προστατικότητα γιατί εδώ δεν πρόκειται για επιλεξιμότητα, πρόκειται για κάτι άλλο. Αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί τελικά. Ε, το επίπεδο ε, κινδύνου. Η πρόθεση να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου που δεν αρνούνται να συμμετάσχουν οι τράπεζες. ε, βεβαίως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο. Αλλά τώρα που δεν ε, λαμβάνονται χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπάρχουν τόσο πολλά ε, προγράμματα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο δια μαγείας. Ε, μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή αυξάνονται στο επίπεδο του κινδύνου. Γιατί τελικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Απενδύσεων δεν πρόκειται να πειραστεί από όλο αυτό. Μάλλον θα μειώσει το λοιπόν, στοιχείο της προστατικότητας και στο στοιχείο του κινδύνου. Όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία τώρα. Ε, έγιναν τεράστιες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα φύγουν ενώ άλλοι δεν ε, πήραν σε άλλες χώρες δεν έγιναν αυτές οι επενδύσεις και μια τελευταία παρατήρηση αφορά το εξής Αυτή τη στιγμή έχουμε ταυτόχρονα διαδικασία με διαδικασία Omnibus. Και αν τη διαβάσετε, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποιες ε, νομικές διατάξεις μέσα των οποίων το ΕΦΣΥ μπορεί να συνθέμει περισσότερα προγράμματα συνοχής. δεν υπήρχε πρόθεση να υπάρξουν ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία να εισρεύσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όχι να ληφθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι, πρόκειται για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ε, και ε, παραπείται η αρχική ιδέα. Πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να μιλούμε για τις ε, προσαρμογές ε, ε, μέσω του Omnibus. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποτελέσει μια διαδικασία, μια κατάσταση win-win εδώ για την δική μας Επιτροπή. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε. Να υπογραμμίσω ότι ο στόχος του ΕΦΣΙ εξ αρχής ήταν η αύξηση των επενδυτικών δυνατοτήτων στην Ένωση. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αν θέλουμε να το πετύχουμε, θα πρέπει να μην υπάρχουν επικαλύψεις με υπάρχοντα άλλα προγράμματα, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις και με την πολιτική συνοχής. Πάντως η αρχική πρόταση ήταν να μην υπάρχει, όπως είπαμε, αυτή η επικάλυψη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα χρηματοδοτήσουμε άμεσα προγράμματα και ε, προγράμματα σε εισαγωγικά οριακά σε επίπεδο κινδύνου. Όχι πολύ ελκυστικά δηλαδή για τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης. Αν δει κανείς τι έχει γίνει μέχρι τώρα, βλέπει ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, σε εισαγωγικά θερμοκοιτίδες ε, παραγωγής προγραμμάτων που βοηθούνται, αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος του ΕΦΣΥ, γιατί εδώ μπλέκεται με τη συνοχή. Και πολλές φορές είναι προγράμματα τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, έχουν μπει στην αρχή αν θέλετε της εκκίνησης, και στο τέλος ελείπουν από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης ε, ε, γιατί τα απορροφά τα ταμεία αυτά το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση συζητάμε το πώς στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να καταθέσουμε δυνατέ τι επενδύσει. Είναι θετικό το, το συζητάμε αυτό, το κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να διευκολύνουμε τι επενδύσει στην Ευρώπη. Μπορούμε φυσικά να τα δούμε όλα μισογεμάτα ή μισοάδια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μισογεμάτο θεωρώ το ποτηρί. Είναι καλό το ότι καθόμαστε και σκεφτόμαστε το πώ θα γίνουν επενδύσει στην Ευρώπη. Αλλά μην είμαστε και αφελεί. ακούγοντα τη σημερινή συζήτηση, Γίνεται σαφές ότι το ΕΦΣΙ αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι φανταζόμαστε στην αρχή και συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Μάλεπτιτς και Φανίστερο ότι φαίνεται λες και το ΕΦΣΙ θα πάρει τα χρήματα από τα αρφαντικά ταμεία και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας φοβίζει. Δεν υπάρχει και αξιολόγηση σωστή στην παρούσα φάση, γιατί έχουμε αποφασίσει πολιτικά, πολιτικός πώς ότι θέλουμε να αυξηθεί αυτό το μέσο. Αλλά μήπως όταν ε, αυξηθεί και άλλο το εύση θα υπάρχει άλλη επικάλυψη με αυτά που κάνουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Ίσως θα πρέπει και εμείς λοιπόν να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τα διαφορετικά κονδύλια να αξιοποιούνται καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς ε, θα είναι πιο απλές οι διαδικασίες μας και επίσης να διευκρινίσουμε ότι κανείς ουσιαστικά στην Ευρώπη δεν ξέρει τι χρηματοδοτείται με τα ευρωδικά ταμεία. Βγείτε στον δρόμο και ρωτήστε κάποιον. Τι χρηματοδοτείται με τα διευθυντικά ταμεία, κανείς δεν ξέρει. Και εδώ θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα marketing, προβολής. Θα πρέπει να πούμε στους ενδιαφερόμενους ότι πρόκειται για χρήματα, κονδύλια, τα οποία έχει νόημα να, αξιοποιηθούν. Φυσικά και υπάρχουν κριτήρια, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, στους πολίτες, τι κάνουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, μπορεί να μα αντικαταστήσει κάποια στιγμή το ΕΦΣΙ και αυτό θα είναι κρίμα και μεγάλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Πούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σας απασχολήσω. Οι συνάδελφοι μας ε, ανέφεραν ε, ποια είναι η κατάσταση, ξέρουμε από πού ερχόμαστε και ποιο ήταν ο σκοπό. Θέλαμε να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσει, αλλά δεν το καταφέραμε και παράλληλα θέλαμε. Θέλουμε πολλά να πετύχουμε. και να κοιτάξουμε τι έγινε και με την, ε, τα Ταμεία Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχουμε ε, μεγάλη εμπειρία και σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν τα χρήματα αυτά να μην αντικαταστήσουν τελικά ε, τα βετικά ταμεία. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για όλα τα κρατημέλη και κυρίως για κρατημέλη από την Ανατολική Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να φροντίσει και για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης σε ό,τι αφορά την πρόσβαση δηλαδή στο πρόγραμμα αυτό γιατί κοιτώντα τον χάρτη των προγραμμάτων αυτών βλέπουμε ότι δεν υπάρχει απορρόφηση στα κρατημέλη αυτά. Δεν υπάρχει επαρκής ε, εκπροσώπηση. Θέλουμε λοιπόν τα κονδύλια. Δεν θέλουμε τα κονδύλια από τα ρευστοτικά ταμεία να καταλήξουν στο ΕΦΣΙ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο, και για τα σχόλια αυτά. Ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι η ευθύνη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι ιδιαίτερη στην παρούσα φάση. Γιατί θα πρέπει να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Σκόπμεϊρ. Η κυρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή και ζωντανή συζήτηση και για την ευκαιρία που μας ε, δίνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο δηλαδή. Και φυσικά σημειώνουμε πάρα πολύ καλά όλα όσα θίξατε στην Επιτροπή σας. Σημειώνουμε και όλα αυτά τα οποία επισημένονται και στο σχέδιο γνωμοδότησης για το ΕΦΣΥ. Η πρόταση θα πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής μέχρι τώρα αλλά και των αξιολογήσεων που έχουν γίνει ως τώρα. Το τονίζω αυτό, γιατί έχουν γίνει αξιολογήσεις ε, τρεις συγκεκριμένα για το ΕΦΣΥ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι δημόσια στοιχεία. Έγινε επίσης ε, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και μία ανεξάρτητη από την Ernst αξιολόγηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν εγκαίρως για να ενταχθούν και στα πλαίσια της συζητήσεις εξ αρχής. Αυτό λοιπόν ήθελα να το πω αυτή εξ αρχής. Τώρα, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε πετύχει έως τώρα. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας τι έχει γίνει τα τελευταία 1,5 χρόνια. Από το τέλος του 2016, το ΕΦΣΥ αναμενόταν να κινητοποιήσει 164 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια επενδύσει σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα μισά, δηλαδή από το 315-315 τα οποία επανεδόν να υπάρξουν ε, σε τριετή περίοδο. Γι' αυτό σε 388.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα θεωρούμε ότι το ΕΦΣΙ έχει πετύχει εν μέρη το στόχο του σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των ενεργητικών κονδυλίων. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολλά, πρόγραμμα, πολλά προγράμματα έχουν ωφελήσει τις ευρωπαϊκές κοινότητες και δήμους, για παράδειγμα στην Ιταλία. Εξυγχρονίστηκε το δίκτυο ηλεκτροδότησης ε, και υδροδότησης ε, στην Πολωνία. Το ΕΕΦΣΙ χρηματοδοτεί 1.300 εγκαιστικές μονάδες στο Πότσναν και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία διατίθονται όλα δημοσίως στο website της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όλα αυτά τα προγράμματα λοιπόν. Να σημειώσω επίσης στο πλαίσιο αυτό το μεγάλο δυναμικό συνδυασμού του ΕΦΣΥ με επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκών Ταμείων. Αυτά είναι συμπληρωματικά και υποστηρίζουν το ένα το άλλο για να επιτύχουν κοινού στόχου. Ποιοι είναι οι κοινοί στόχοι, μεγαλύτερε επενδύσει, οικονομική ανάπτυξη, θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με χαρά σα ανακοινώνω ότι έχουμε δει επιτυχή παραδείγματα τέτοιων συνδυασμών ω τώρα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα. Τα Νοχπακαλέ, ένα project που προωθεί την οικονομία χαμηλού, χαμηλών εκπομπών ανθρακάν. Η Γαλλική Τράπεζα, οι ιδιωτικοί επενδυτέ εμπλέκονται μεταξύ άλλων. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάκουσε τις κριτικές που ακούστηκαν για το ΕΦΣΥ και για τη λειτουργία του Ταμείου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς αυτές τις κριτικές φωνές θέλει να απαντήσει. Και πώς? Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η πρόταση βασίζεται στην εφαρμογή του ΕΦΣΙ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Μεγάλο στοιχείο και μεγάλο κομμάτι του, της πρότασης για το ΕΦΣΙ. Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε τεχνική αρρωγή σε τοπικό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδύσεων και αυτός ο κόμβος προβλέπεται ότι ενεργά θα πρέπει να συμβάλλει στους στόχους και της τομεακής αλλά και της περιφερειακής διαφοροποίησης του ΕΦΣΥ στη φάση της εφαρμογής αλλά και της προετοιμασίας. Ο κόμβος να σας πούμε ότι ήδη για κάποια project έχει τεθεί σε λειτουργία αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τοπικές ε, ικανότητες και ιδιαίτερα σε συνεργασία με τις ε, περιφερειακές και εθνικές τράπεζες, όπου αυτό χρειάζεται πιο πολύ προφανώς. Επίσης προτείναμε μεγαλύτερη υποστήριξη για τις ε, πλατφόρμες επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και τις μεταβατικές περιοχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διαβρινθεί η τομεακή κάλυψη με αναφορά σε οποιαδήποτε κλάδο που δεν θα καλύπτονταν ιδάλλως στους γενικούς στόχους του ΕΦΣΗ. Να αναφερθεί η γεωργία, η αλία, οι δατοκαλλιέργειες ως ε, ρητή που μπορεί να καλύπτονται από το ΕΦΣΗ. Επίσης, τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αποφευθεί η υποστήριξη των αυτοκινητοδρόμων όπως αναφέρθηκε σήμερα. Εκτός αν αυτή η υποστήριξη χρειάζεται για να υποστηριχθούν οι ιδιωτικέ επενδύσεις στις χώρες του Ταμείου Συνοχής. Ένα άλλο βασικό θέμα το οποίο θα θέλαμε να υπογραμμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η συμπληρωματικότητα. Βασικό στοιχείο του ΕΦΣΥ προτείνουμε να ξεκαθαρίσει ακόμα πιο πολύ ότι τα προγράμματα θα πρέπει να δίνουν μία απάντηση σε κενά που υπάρχουν στην αγορά. Και αυτό να περιλαμβάνεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και πιο σαφή ορισμό τη συμπληρωματικότητα προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο ακριβή κριτήρια δηλαδή για το τι θεωρείται συμπληρωματικό. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να θερούνται εκ των προτέρων συμπληρωματικά τα δυσνοριακά έργα, δεδομένης της σημασίας που έχουν και της δυσκολίας που υπάρχει στην πρόθεση αυτών και στην εφαρμογή τους. Διαφάνεια, άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε και σήμερα, θα ενισχυθεί περαιτέρω. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι η Επενδυτική Επιτροπή που περιλαμβάνει τους ε, εμπειρογνώμονες να λαμβάνει αποφάσεις για τη χρήση των εγγύησεων. Αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε την Επιτροπή ούτε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, ότι η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να εξηγεί λεπτομερώς και εντελεχώς γιατί επιλέχθηκε το κάθε έργο και πώς πληρούνται τα κριτήρια για να αποδεχθεί ακριβώς ο συμπληρωματικός χαρακτήρας. Να σας πω ότι υπάρχει συνδυασμός του ΕΦΣΥ με άλλα ταμεία, τα δοσοτικά ταμεία ω επιτοπλίστων. Αυτό αποτελεί βασικό στόχο της πρότασης ΕΦΣΥ 2, το οποίο περιλαμβάνεται και σε μια συμπληρωματική πρότασία Omnibus που α, τροποποιεί τον ε, εφαρμοστικό κανονισμό και αυτό θα αφορά και τις πλατφόρμες επενδύσεων αλλά και τα μεμονωμένα έργα. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η δημιουργία πλατφόρμων επενδύσεων, είτε είναι σε εθνικό, διασυνοριακό επίπεδο κτλ., θα συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους Δήμους και τις κοινότητες. Έχουμε δει να δημιουργούνται τέτοιες πλατφόρμες και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Και κλείνω με την ελπίδα ότι μετά την έγκριση από πλευρά του ΕΚΟΦΗΝ για το FC 2.0 πέρσι το Δεκέμβριο, ούτε τρει μήνε δεν έχουν περάσει δηλαδή. Δεν πέρασαν από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να πάμε για λίγο πιο γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο πριν το θερινό διάλειμμα. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Συγγνώμη που σα κούρασα. Γεια σα. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπρέσο, θέλετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν οι συνάδελφοι. Δεν είναι όλες ε, οι παρατηρήσεις που έγιναν αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Ανήκουν περισσότερο στην, ε, στον προϋπολογισμό και στις άλλες επί της ουσίας αρμόδιες επιτροπές. Αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε επίπεδο οικονομικό αν θέλετε. Συγγνώμη για το τηλέφωνό μου, αλλά χτυπάνε συνέχεια γύρω από την έκθεση αυτή. Θα το κλείσω. Λοιπόν, θα ήθελα σαν οικονομολόγος να πω κάτι. Το ΕΦΣΥ, αν μπορεί να το πει κανείς, ήταν το πρώτο μέσο το οποίο έδωσε στον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις, αν και χρηματοδοτήθηκαν εκ των υστέρων και τέτοιου είδους. Εκτός των διαφθορωτικών ταμείων, τα οποία στην αρχή είχαν σαν βασικό στόχο να συγκλίνουν οι οικονομίες. ή κάλυπταν κάποιες περιφέρειες αναπτυγμένων χωρών σε κρίση. Μετά υπήρξε, ξέρετε, μία μεταρρύθμιση των κανονισμών των διαφορετικών ταμείων και αυτό οδήγησε ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες περιοχές να υπάρξει καλύτερη δυνατότητα στήριξη των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Πάντα όμως παραμένουμε στα πλαίσια ενός προσανατολισμού με βασικό στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης. Ε, μέσω του ΕΦΣΥ για πρώτη φορά και παραδεχτήκαμε για πρώτη φορά ότι η πολιτική του όχι στις κρατικές παρεμβάσεις όταν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, από την Κίνα μέχρι τις, Πολιτείες, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. παντού υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις. Η στάση δική μας δεν ήταν η καλή και έγινε λοιπόν μια πρώτη πρόταση, ανεπαρκής ίσως, υποστήριξη των επενδύσεων, κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων, έτσι ώστε να επιτρέψουμε σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης να αναλάβουν συγκεκριμένους κινδύνους γιατί η ανάγκη αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στην Ευρώπη για την αύξηση των επενδύσεων. Οι επενδύσεις στην Ευρώπη μετά από την οικονομική κρίση είχαν συντριβεί και το ΕΦΣΥ μπόρεσε ε, έστω και επιμέρους να καλύψει εν μέρη το κενό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε αναζητώντας το καλύτερο να μην αποτύχουμε στο καλό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τις επενδύσεις, όχι μόνο τις δημόσιες, αλλά και τις ιδιωτικές. Το πρόβλημα δεν είναι να πούμε εμείς, ας καταργήσουμε τα εύση και από εκεί και πέρα ας βολευτούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Δυστυχώς αυτό από μόνο του δεν ισχύει. Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν θα στηρίξουν την αγορά μόνες τους. Και πρέπει να προσέξουμε να βελτιώσουμε το μέσο αυτό. Δεν έχουμε άλλο στη διάθεσή μας τον τομέα αυτό και να διευρύνουμε τις δυνατότητες επιρροής του ΕΦΣΙ στην πραγματική οικονομία. Κάτι τέτοιο ε, θα έλεγα ισχύει κυρίως για κλάδους της οικονομίας οι οποίοι ακόμα δεν μπόρεσαν να καλυφθούν από το ΕΦΣΙ. Πρέπει λοιπόν μέσω της τεχνικής ε, αρρωγής και μέσω των ε, εθνικών πόλων συμβούλων να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επενδύσεις και δεν αναφέρομαι τόσο σε δημόσιες επενδύσεις όσο σε ιδιωτικές. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν εξοικονομούν πολύ, αλλά αυτό δεν μετατρέπεται σε κονδύλια επενδυτικά. Το να δοθούν λοιπόν κάποιες εγγυήσει για τους κινδύνους τους οποίους πρέπει να αναλάβουν οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι στόχος βασικός για την Ευρώπη. Θα πρέπει να προσανατολίσουμε λοιπόν την κριτική μας, όχι λέγοντας ότι δεν είναι χρήσιμο το εύση, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να χρησιμεύσει με καλύτερο τρόπο από ό,τι τώρα και πώς θα καλύψουμε τα προβλήματα τα οποία πράγματι έχουν εντοπιστεί. Αυτό είναι ο στόχος τον οποίο εγώ σας προτείνω. Εμείς δεν μπορούμε να διαγράψουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να βοηθηθεί η Ευρώπη στις επενδύσεις της. Εμείς θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είμαστε η Επιτροπή η οποία φέρνει σε επαφή, αν θέλετε, τις πιο πλούσιες οικονομίες της Ευρώπης με τις λιγότερο πλούσιες. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι οικονομίες που δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το ΕΦΣΙ για τον ιδιωτικό τους τομέα να το κάνουν. Αυτό θα το κάνουμε εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους πόλους, σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πρώτον, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν θέλουμε με εθνικέ ποσοστώσεις, αλλά θέλουμε μια γεωγραφική ισορροπία, σταδιακά επιτεύξιμη και ταυτόχρονα μέσω και της άμεσης, ε, αν θέλετε, επιχορήγησης, η εμπειρία μας δείχνει ότι δεν πρέπει να ονομάζουμε μόνο τα πράγματα και να μένουμε στα λόγια, αλλά να βοηθάμε, να βοηθάμε και στη σχεδίαση και στην δημιουργία δομών ενδιαμέσων στις διάφορες χώρες, όπως οι εθνικές πλατφόρμες, η εθνική πόλη. Ε, είναι σημαντικότατη γιατί έτσι θα επιτρέψουν να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα προγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για τα δημεθοριακά προγράμματα, τα οποία είναι για μένα κυρίαρχή σημασίας. Δύο επιμέρους απαντήσεις έτσι ώστε ε, να συζητήσουμε τα θέματα αυτά εκ νέου στο μέλλον. Εγώ θυμίζω ότι παραμένω στις αρμοδιότητές μας, γιατί αν φύγουμε από τις αρμοδιότητές μας, ή επί της ουσίας επιτροπές ε, θα μας πούν ότι μην ασχολείστε με τα θέματα αυτά, είναι δική μας υπόθεση, όπως το κάνουμε και εμείς όταν μας δίνουν γνωμοδοτήσεις οι οποίες δεν είναι σχετικές. Γύρω λοιπόν τώρα από τις τροπολογίες τις οποίες ήδη έχω παρουσιάσει υπήρξαν ορισμένες ερωτήσεις για, από τους συναδέλφους. Για την τρία, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι θα ήταν λάθος να περιοριστούμε στις ε, φυσικές, αν θέλετε, υποδομές και τις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει να μιλάμε για τέτοιου είδους ε, ε, υποδομές, αλλά και μία πτέσα. Ε, υποδομές όπως σαν παραδείγμα η έρευνα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και είναι και πιο σημαντικό από τις απτές πραγματικές υλικέ μορφές επένδυσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει ε, να μιλήσουμε για το συντονισμό ανάμεσα σε περισσότερες από μία ή δύο χώρες. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο διαμεθοριακός και νομίζω ότι καλύπτω εδώ τους συναδέλφους σχετικά τώρα με την τροπολογία υπαριθμών 10. Ακριβώς και γιατί πιστεύω ότι η χρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για τις χώρες συνοχής θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ακριβώς όταν τίθενται θέματα όπως η ικανότητα της αγοράς να καλύψει το κόστος ή δεν τίθεται σε εφαρμογή η αρχή της προσθετικότητας και δεν αρκούν τα διαφθορωτικά ταμεία. Το θέμα δεν είναι λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε να αποδυναμώσουμε τα διαφορετικά ταμεία, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και αυτά εκεί όπου υπάρχουν στοιχεία αποτυχίας της αγοράς ή υπάρχει έλλειψη αποδείξιμης προσθετικότητας, διότι όπως αρκετοί έχουν ήδη επιθυμήσει, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε τον σημαντικότατο ρόλο των διαφορετικών ταμείων. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε για το ότι το ΕΦΣΙ δεν είναι το υποκατάστατο των διαφορετικών ταμείων. Το διαφορετικό ταμείο, τα διαφορετικά ταμεία έχουν άλλους στόχους και για την χρηματοδότηση των περιφερειακών πολιτικών, όχι προγραμμάτων μόνο, και δεύτερον τα περισσότερα από τα διαφορετικά ταμεία έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τις επιμέρους περιφέρειες που υστερούν προς αυτές οι οποίες είναι πλουσιότερες διασφαλίζοντας την ανάπτυξή τους. Και γι' αυτό λοιπόν εξυπηρετούν πολιτικές και όχι μεμονωμένα προγράμματα. Καμία λοιπόν περιφέρεια δεν έχει βοηθηθεί σε επίπεδο διαφθρωτικό σε ε, μεμονωμένα προγράμματα. Λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει εμείς να μην ε, υποκύψουμε στην πρόκληση να χρησιμοποιήσουμε το ΕΦΣΥ για πολιτικές οι οποίες ε, δεν είναι αυτές που πρέπει να ακολουθήσουμε και να στηρίξουμε όπως οι πολιτικές συνοχής οι οποίες ανήκουν στην πολιτική της συνοχής. Λοιπόν, συμφωνούμε πάνω κάτω. Η μάχη δεν δίδεται σήμερα. Σήμερα συζητάμε για την εξέλιξη του ΕΕΣΥ και το πώς θα αυξήσει την ικανότητά του εξυπηρέτησης των πολιτικών συνοχής και όχι μόνο των γενικότερων επενδυτικών πολιτικών, προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας κονδύλια από τις πολιτικές συνοχές. Αυτό είναι το ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να στείλουμε. Εμείς νομίζουμε, θεωρούμε ότι το ΕΦΣΙ και τα διαφορετικά ταμεία μπορούν να συνεργάζονται, όχι αποδυναμώνοντας το ένα το άλλο, ενισχύοντας τα διαφορετικά ταμεία, τα οποία μερικές φορές δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των ιδιωτικών επενδύσεων. Γιατί με τα διαφορετικά ταμεία δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λοιπόν ένα πρόγραμμα επενδύσεων ιδιωτικό, το οποίο να είναι συγκλίνων με άλλα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα, μέσω του ΕΦΣΥ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους και από κοινού τα ταμεία αυτά να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις συγκλήσεις ανάμεσα στα δύο αυτά τα μία και όχι να υποκαταστήσουμε το ένα με το άλλο. Τουλάχιστον αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας στο μέλλον. Θα δούμε πώς θα πάνε οι επενδύσεις μας. Το μήνυμα όμως το οποίο θα πρέπει να στείλουμε και το οποίο υπάρχει στο γραπτό κομμάτι του κειμένου είναι σαφές. Η πρόεδρος μου λέει να μην μακρηγορώ δίκιο έχει αλλά θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό όταν εξετάσουμε συγκεκριμένα τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά ήταν κάπως ε, πιο μακροσκελής από ό,τι περιμέναμε. Θα ήθελα να υπέθυμίσω σε όλους ότι η μερμηνία για την κατάθεση ε, τροπολογιών είναι το μεσημέρι της Δευτέρας ε, της δεκάτης ε, ε, της, 30, ε, 30 Ιανουαρίου συγγνώμη. τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπούντα για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της προβολής της επιδόσης των Ευρωπαϊκών Διαφορετικών και Επενδυτικών ε, Ταμείων. Αυτό είναι το θέμα του. Και έχετε το λόγο, κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω <clears throat> ευχαριστώντας όλους τους ε, συναδέλφους, γιατί ε, κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να εκπονηθεί μια έκθεση αυτού του τύπου. Ευχαριστώ πολύ ε, ε, όλους και ιδιαίτερα στον κύριο Λάμπερτ. Είναι σημαντικό ότι στο τέλος αυτή τη έκθεση να γνωρίζονται νέοι μέθοδοι, ούτω ώστε να έχουμε μια ενισχυμένη ε, πολιτική συνοχής, ούτω ώστε η πολιτική αυτή να διαδραματίσει ένα πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, έχουμε ανάγκη μιας ισχυρής οικονομικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει εδώ μια άλλη λεξάρτηση και τα δύο βεβαίως εξαρτώνται και από την πολιτική συνοχή. Υπήρξε μια άξη των επενδύσεων πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ χάρη ακριβώς στην πολιτική συνοχή. Αυτό εκπροσωπεί μια αύξηση πάνω από 60% επενδύσεων σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένες χώρες η αύξηση των επενδύσεων ανήλθε μέχρι τα 80%. Και όλα αυτά οφείλονται στην πολιτική της συνοχής. Η πολιτική αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο επιτρέπει να διοχετεύουμε τα κονδύλια προς τις πιο φτωχές ε, περιοχές. Και ταυτόχρονα η πολιτική αυτή επιτρέπει να μειώσουμε τις διαφορές, να βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών. Η πολιτική χρηματοδότησης οι πολιτικές μάλλον χρηματοδότηση έχουν πάντοτε μια θετική επίπτωση στους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Συχνά η καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών άλλαξε ριζικά ακριβώς ε, χάρη στον επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Δυστυχώς οι επενδύσεις αυτές δεν κατανέμονται με δίκαιο τρόπο και το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι μόνο ένα μικρό κλάσμα Ευρωπαίων πολιτών έχουν συνείδηση ε, των ε, ευρωπαϊκών επιπτώσεων των επενδύσεων στην ε, περιφέρειά τους. Κατά συνέπεια, στην έκθεση αυτή οι ιδέες πρωτοβουλίας προσπάθησα να δω πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να μιλήσουμε για πραγματικές απτές και θα θέλαμε επίσης να αναφερθούμε στη διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ πολιτικής συνοχής από τη μία και των οργάνων, των εργαλείων της ε, τοπικής ε, περιφερειακής πολιτικής ε, πώς ε, μπορούμε να καταστήσουμε υποτελεσματική την περιφερειακή πολιτική και να αυξήσουμε το επίπεδο συμμετοχής των, ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε να προβάλλουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των ε, κονδυλίων, ούτως ώστε να μιλήσουμε για την προσθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής. Πώς μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική χρησιμοποιώντας επί παραδείγματι κοινωνικά δίκτυα, τις online πλατφόρμες. Πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ευθύνη, την κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Και υπογραμμίζω, μπορούμε να το πράξουμε εφόσον όλοι οι εταίροι που ενέχονται σε όλες τις ε, φάσεις εφαρμογής μπορούν να συμμετάσχουν. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να μείνουμε στο γεγονό ότι ε, αυτοί που επεφελούνται από τα ταμεία θα πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικούς πρέσβεις της ε, πολιτικής ε, συνοχής, ούτως ώστε να μιλήσουν αποτελεσματικά για τα ευεργετικά ωφέλη της πολιτικής αυτής και θέλουμε να εντοπίσουμε κάποιους ε, τρόπους ούτως ώστε να επιτρέψουμε στους πολίτες να συμμετάσχουν περισσότερο σε όλες τις ε, δημόσιες διαβουλεύσεις και να είναι πιο παρόντες σε όλα τα δίκτυα που επιτρέπουν την καλύτερη διάχυση των πληροφοριών. Και θα ήθελα να ε, μοιράσω την έκθεση σε δύο τμήματα. Καταρχήν μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία και δεύτερον το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ενεχόμενων μωρών στην ε, διαδικασία διαβούλευση και στην ε, εφαρμογή. Για το πρώτο τμήμα, μια καλύτερη επικοινωνία, πώς να αγγιθούμε μεγαλύτερη ορατότητα για την, ε, στην πολιτική συνοχή; Στην Επιτροπή μας, κατά επανάληψη είπαμε, ότι θα πρέπει η νομοθεσία να απλουστευτεί. Πολλές χώρες μέλη λυπούνται για το γεγονός ότι οι διαδικασίες είναι υπερβολικά περίπλοκες όσον αφορά τα χρήματα τα οποία εκταμιεύονται από αυτά τα ταμεία. Οι εθνικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να υιοθετήσουν κάποιες ε, εθνικές στρατηγικές ε, ούτως ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση οι περιφέρειες των εν λόγω χωρών. Οι αρχές διαχείρισης έχουν το καθήκον να χρησιμοποιήσουν πιο προσαρμοσμένα στο σκοπό αυτό εργαλεία. Είναι σημαντικό να δούμε πώς οι εθνικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να δραματίσουν ένα πιο καθοριστικό ρόλο. Γιατί με τον τρόπο αυτό η γρατότητα της πολιτικής αυτής ε, στα μάτια των πολιτών θα αυξηθεί. Και ένα άλλο θέμα. Ε, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα τη θετική αξία των ε, αποτελεσμάτων μας. Θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση ευρωπαϊκής επικοινωνίας, ούτως ώστε να μπορούν να διαβάζονται συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία να είναι πιο εύληπτα για τον Ευρωπαίο πολίτη, ώστε να υπογραμμίσουμε ποιε είναι οι σορευθήσεις εμπειρίες και τα αποτελέσματα και αναφέρομαι στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθησαν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ότι δεν ε, χρειάστηκε καν στις περιπτώσεις αυτές να υπάρξει μια δημοσιοποίηση, μια κοινοποίηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι, αυτή είναι βαρύτατη αμέλεια. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα πρέπει να επικοινωνεί καλύτερα τα θετικά του αποτελέσματα και οι Ευρωπαίοι πολίτες καμιά φορά δεν έχουν πρόσβαση στις ε, πληροφορίες αυτές. Πράγμα που είναι λυπηρό. Μόνο 9% των πολιτών που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου γνώριζαν ότι κάποια προγράμματα είχαν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι υπερψήφισαν το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σε περιφέρειες όπου είχαν αξιοποιηθεί περισσότερο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό αποτελεί παράδοξο και πραγματικά είναι και κρίμα όσον αφορά τις εξελίξεις. Στην Πολωνία το ποσό των πολιτών που γνωρίζουν ότι στην περιφέρειά του χρηματοδοτούνται κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίση περιορισμένο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μόνο ε, μέσο επικοινωνίας. Και υπογραμμίζω, υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της ε, ψηφιακής ε, επανάστασης, ψηφιακής εξέλιξης ότι θα διευκολύνουμε την επικοινωνία, την ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, υποθελούμενων από τα προγράμματα και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Να υπάρχει μια ηλεκτρονική επικοινωνία. Γιατί με τα ηλεκτρονικά μέσα μπορούμε να επισημάνουμε τα προβλήματα και να βρούμε μια ταχεία λύση. Και τώρα θα περάσω στο δεύτερο τμήμα της έκθεσής μου. Έλεγα ότι θα πρέπει να ανθαρρύνουμε τη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μοντέλα συνεργατικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει δηλαδή να επιτραπεί στους τοπικούς ε, φορείς και παράγοντες να χρησιμοποιήσουν έναν ε, συνεργατικό προπολογισμό. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να εντοπίσουμε τα εργαλεία τα οποία θα επέτρεπαν στις ε, τοπικές αρχές να αυξήσουν το βαθμό συνεργασίας τους σε όλες τις διαδικασίες πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα θέλαμε να έχουμε ένα μέγιστο αριθμό πολιτών που να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων. Όσον αφορά τώρα την ε, αναβάθμιση του ρόλου των εταίρων, ε, στην ε, συγκυρία ακριβώς δημιουργίας εταιρικών σχέσεων. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι θεμελιώδες για τις εταιρικές επενδύσεις, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδο θα πρέπει να αντιλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν. Αύξηση της ε, περιφερειακής συμμετοχής θα αγγελθεί καλύτερα αποτελέσματα επί τόπου. Και ε, αν δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, αυτό θα προπέθεται μια στενή συνεργασία μεταξύ ε, αστικών, δηλαδή υπηρεσιών που αφορούν τις αστικές περιοχές και την Ήπεθρο ακριβώς όπως και τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Η συνέργεια των ταμείων έχει ήδη αναφερθεί και εγώ η ίδια πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντική. Και θα ήθελα να κλείσω εδώ αναμένοντας με ανυπομονησία τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Και θα ήθελα τελικά να έχουμε μια καλή έκθεση για να τονίσουμε τον καθοριστικό ρόλο της πολιτικής ε, συνοχής. Σας ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το Μάρτιο θα γίνει η παρουσίαση του θέματος και η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το Μάιο. Οι συντονιστές τώρα. Να είστε παρακαλώ σύντομοι. γιατί ήδη περιμένει απ' έξω ο επόμενος ομιλητής, ο επόμενος προσκεκλημένος μας από την ε, Προεδρία της ΜΑΝΤΑΣ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ξεκινήσω όμως υπογραμμίζοντας ότι το θέμα μη εξασθένησης της ε, των διαφορετικών πολιτικών αποκτά τη διάσταση που της αρμόζει και προκαλεί το ενδιαφέρον που απαιτείται. Νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε ε, τι σημαίνει η Ευρώπη για τους πολίτες, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει το τι δεν πάει καλά. Το 1 τρίτο του προϋπολογισμού πηγαίνει στην πολιτική συνοχή και οι πολίτες δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει ένα τεράστιο ρήγμα το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ε, που συνδυάζει τα ερευνητικά Ινστιτούτα, τα κέντρα επικοινωνίας κτλ. θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει μία πρόταση για τη σχέση της έρευνας με τις επενδύσεις. Πάντως τα αποτελέσματα θα μας γνωστοποιηθούν στο τέλος. Έχουμε στη διάθεσή μας μόνο επιμέρους στοιχεία, πάντως τα οποία λέγουν ότι τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υπόθεση του roaming. Ε, της, ε, αυτής της δραστηριότητας λοιπόν είναι κάτι το οποίο οι πολίτες των Ευρωπαίων πολιτών δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ε, σημασία. Ιδιαίτερα το 1 τρίτο των πολιτών της Ένωσης που αλλάζουν συχνά ε, χώρες. Συνεπώς λοιπόν μια τόσο σημαντική αν θέλετε διαδικασία σε αυτή της περιαγωγής ε, είναι απαράδεκτο να μην είναι γνωστή και να μην είναι γνωστοί οι λόγοι ε, για τους οποίους ε, δεν ε, είναι γνωστή η δραστηριότητα αυτή. Από αυτά τα οποία λέγει ο κύριος Μπούντα, μας δείχνει ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να γίνεται κατανοητή μόνο από το 25% των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό δεν είναι επαρκές και μάλιστα είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, του πληθυσμού, το οποίο ταξιδεύει συχνά και το οποίο μιλεί ξένες γλώσσες. Το θέμα λοιπόν είναι ποιος θα διαφημίζει, αν θέλετε, την πολιτική της συνοχής. Τα μέσα μπορεί να είναι πολλαπλά, αλλά σε τοπικό επίπεδο η, ε, αν θέλετε, παρουσίαση των προϊόντων αυτών, των επενδυτικών, θα πρέπει να γίνεται από τις τοπικές αρχές οι διαχειριστικές αρχές και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να κάνουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε διαφορετικούς τομείς και με διαφορετικούς στόχους. Ε, να γνωρίζουν οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το πώς μπορεί να συμμετέχουν στα προγράμματα, το πώς μπορεί να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό και αυτό θα πρέπει να γίνεται όχι στις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει να γίνεται επί τόπου. Θα πρέπει επίσης όλα αυτά να γίνονται με κυκλική, αν θέλετε, μορφή, έτσι ώστε η ενημέρωση του κοινού να παραμένει σταθερή. Νομίζω ότι έτσι και θα ενημερώνουμε, αν θέλετε, τους θεατές σε εισαγωγικά, τους πολίτες που δεν συμμετέχουν, αλλά θα διευκολύνουμε ταυτόχρονα και την δυνατότητα παρέμβασης των εμπλεκομένων, δηλαδή επιχειρηματιών και τοπικών αρχών κτλ. Αυτό δεν σημαίνει τοπικές, ότι οι τοπικές αρχές ή μάλλον σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρητικά έχει μια ευρύτατη εικόνα για το τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Οι πλέον βέλτιστες των πρακτικών θα πρέπει να γνωστοποιούνται ε, και να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε θέματα όπως ο γεωεντοπισμός, το geolocalization και ταυτόχρονα να καταστήσουμε πραγματικούς εταίρους και τις πιο απομεμακρυσμένες περιοχές ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας που υπάρχουν. Ε, ένας άλλος τομέας τον οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η επικοινωνία ανάμεσα στις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές. Θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, περισσότερη ενημέρωση για τα κονδύλια τα οποία προέρχονται από την Ευρώπη και χρησιμοποιούνται. Ε, η ενημέρωση που γίνεται από τις εφημερίδες είναι με πολύ γενικό τρόπο και καλύπτονται συγκεκριμένοι τομείς και δεν δίδονται, αν θέλετε, δεν δίδεται σημασία στην πραγματοποίηση άλλου είδους, ε, στην ολοκλήρωση άλλου είδους υποδομών. Αυτό δημιουργεί ένα κενό ενημέρωση στους πολίτες, γιατί οι πολίτες ακριβώς ε, καλούνται ε, να γνωρίσουν τι ακριβώς γίνεται με τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται λοιπόν πιο συγκροτημένες παρεμβάσεις έτσι ώστε να κατανοούν οι πολίτες τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα μπορέσουμε, θα έλεγα, να βελτιώσουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε ε, και τα μεμονωμένα προγράμματα και εδώ θα πρέπει ο διαφθρωτικός διάλογος με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα αν θέλετε Κοιτάξτε, καιρό είναι να τελειώσετε, λέει η πρόεδρος. Ε, κύριε Τζουφρίντα λέει ότι είναι απαραίτητο στον τομέα της συνεργασίας ανάμεσα στους τοπικές, στις τοπικές αρχές και τους εμπλεκομένους οικονομικούς εταίρους να βελτιωθεί η συνεργασία τους και να καλύπτουν έτσι με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των εδαφών τους. Λυπάμαι που σας διακόψα, αλλά δεν έχουμε καθόλου ε, χρόνο. Ο κύριος Βανότεμπομ. Θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ σύντομο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε την ε, συζήτηση όταν θα λάβουμε και το σχέδιο της έκθεσης. Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι και η Επιτροπή των Περιφερειών και πολλές τοπικές περιφερειές ε, θα έχουν ιδέες για την ε, βέλτιστη εφαρμογή. Ίσως θα μπορούσαν να ληφθούν λοιπόν υπόψη και να συμμετάσχουν και αυτές, όπως νομίζετε ότι θα πρέπει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να συμπεριληφθούν αυτά στην πρόθεση σας κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ για το ότι ήσασταν και πολύ σύντομο. Η κυρία Βάνα έχει το λόγο. Σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Δεν θα επαναλάβω ε, τα όσα ήδη υπόθηκαν για την προβολή του θέματος. Θα μιλήσω όμως πιο πολύ για την ε, μεγαλύτερη εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Ε, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και για τους ε, κοινωνικούς εταίρους και για την κοινωνία των πολιτών. Γιατί θεωρούμε ότι μόνο με την καλή συμμετοχή της ε, ε κοινωνίας των πολιτών μπορεί να υπάρχει πιο σωστή και πιο καλή εφαρμογή, πιο σωστά αποτελέσματα. Αυτό μας συμφέρει όλους, πιστεύω. Και έχει αποδειχτεί ότι εκεί που έχει συμπεριληφθεί η πολιτική η κοινωνία των πολιτών για θέματα αισότητας, περιβάλλοντος, αποκλεισμού. Εκεί πραγματικά υπάρχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι στην εφαρμογή της αρχής εταιρικής σχέσης υπάρχουν πολλές διαφορές και πολλές χώρες πρέπει να καλύψουν πολύ καμένο έδαφος και πολύ λυπάμαι που αναφέρω ότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Θα πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν αυτή η αρχή σε τοπικό επίπεδο. Θα κάνουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις για έναν κώδικα συμπεριφορά με κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές αλλά και ένα μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για να υπάρχει πραγματική συνεργασία και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Νταμάτο. Έχετε το λόγο για λίγο όμως. Ε, πρόεδρε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στην ε, πολιτική αυτή για να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία και να προβληθούν σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα α, σημείο το οποίο δεν χωράει αμφιβολία. Για μας ιδιαίτερα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να Πρέπει μάλλον να παρατηρήσουμε ότι δεν καταφέρνουμε να περάσουν οι πληροφορίε και η ενημέρωση για την χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε θέματα συνοχή. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο και δεν το καταλαβαίνει ο πολίτη. Και το πιο κλασικό είναι το θέμα της γραφειοκρατίας, ε, ότι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και κρατών μελών. Δημοσιεύθηκε μια έκθεση από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο και αναφέρεται ότι από εδώ προκύπτουν ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης, το 1 τρίτο όλων των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργούνται δηλαδή. Για τι θέσεις όμως μιλάμε. Τι είδους λοιπόν θέσεις εργασίας ε, πρέπει να δώσουμε στους πολίτες μας. Θα πρέπει να είναι πολύ σωστά στοχευμένη η παρέμβαση. Θα πρέπει επίσης η εμπλοκή των εθνικών και των τοπικών αρχών να είναι μεγαλύτερη και ποιοτικότερη και θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή όταν πρέπει να κατηγορήσουν τις Βρυξέλλες για τις ανικανότητές τους τις διοικητικές, που κάτι το οποίο έχει συνέπειες για τις μεμονωμένες χώρες. Τώρα για την αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου, αν θέλετε, σταθερότητας και για την μακροαιρεσιμότητα, εμείς από την αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου λέγουμε ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιους τομείς στον υπολογισμό του χρέους. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σταματήσουμε στο σημείο αυτό τη συζήτησή μας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας τελείωσε. Οι συνάδελφοι που ήθελαν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ να θυμηθούν τι ήθελα να πούν όταν θα κάνουμε την κανονική συζήτηση στην παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης το Μάρτιο. Το Μάρτιο λέω. Και τώρα να καλέσω like to να προσκαλέσω λοιπόν τους εκπροσώπους της Μαλτέζικης Προεδρίας που θα μας παρουσιάσουν τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά τον τομέα αρμοδιότητας των Επιτροπής μας, ε, ο κύριος Γιάνν Μπόρκ, κοινοβουλευτικής γραμματέας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία και για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στη Μάλτα, που θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας Στου τομεί που είναι αρμόδιοι η Επιτροπή μας. Ο θα μας κάνει μια παρουσίαση 15 λεπτών στην πρώτη φάση και μετά θα πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής, καταρχάς οι συντονιστές. Thank you. Thank you very much. So I began with uh, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε το λόγο για την παρουσίασή σας, των προτεραιοτήτων σας και μετά θα έχουμε το γύρο έρωτα απαντήσεων από τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχετε το λόγο κύριε Μπόρκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ και για την επανεκλογή σας ως πρόεδρος της Επιτροπής Επιτροπής Ανάπτυξης. Με μεγάλη χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας σήμερα. Θα είμαι σύντομο ε, στην ε, παρουσίασή μου σε ό,τι αφορά την αξιολόγησή μας για το τι είναι ε, σχετικό στον τομέα αυτό και τι είναι σημαντικό στον τομέα αυτό για τους Ευρωπαίους πολίτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με μέρα και των ασώσεων συμβαίνουν σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τι βασικέ προτεραιότητε τη Μαλτέζικη Προεδρία για του επόμενου 6 μήνε. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σα ε, σχόλια και παρατηρήσει σε ό,τι αφορά τι τρέχουσε προκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του συνολικού στόχου στον τομέα τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις ε, φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχει μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Διάφορες ε, περιστάσεις και διάφορα περιστατικά έχουν ε, προκαλέσει τραύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρομοκρατία, ε, μετανάστευση, τα μεταναστευτικά κύματα και επίσης η απόφαση που ελέγχθησε από την Βρετανία για τον Brexit. Επίσης υπάρχει έλλειψη σταθερότητας στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από την, ε, την ε, αβεβαιότητα που υπάρχει για τις σχέσεις με τους διεθνείς εταίρους. Επιπροσθέτως ε, θα αντιμετωπίσουμε και άλλα ζητήματα φέτος. Έχουμε τις επερχόμενες εκλογές στην Ολλανδία, στην Γαλλία, στη Γερμανία που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις, ε, τις μελλοντικές προτεραιότητες της Ένωσης. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτές δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την ε, συνέχιση της ευρωπαϊκής ατζέντα. Θεωρώ ότι αποτελούν μάλιστα και μια ευκαιρία, να σας πω, για να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη, η οποία θα είναι και πιο ανταγωνιστική και πιο κοινωνική. Ως Προεδρία λοιπόν τονίζουμε αυτή την κοινωνική πτυχή. Η Μάλτα θεωρεί ότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στις αβεβαιότητες. Και γι' αυτό λοιπόν στην Προεδρία μας ακριβώς σε αυτές τις ε, σε αυτούς τους φόβους θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε των πολιτών. Και να σας... Ε, θα θέλαμε πραγματικά να δώσουμε μια απάντηση σε όλα αυτά που απογοητεύουν τους πολίτες. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε λίγο πολύ τις προτεραιότητές μας, τις οποίες και θα αναφέρω στην συντομία, αλλά να σας αναφέρω ότι σίγουρα θα επικεντρωθούμε και έχουμε επικεντρωθεί σε θέματα μετανάστευσης, γιατί και ως χώρα είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι με τα ζητήματα αυτά. Και ως Προεδρία θα θέλαμε να πούμε, το είπαμε άλλωστε και στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα, το διευκρίνησε ο Πρωθυπουργό μας, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφές. Είναι σαφή σε ό,τι αφορά την ατζέντα της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης. Άρα η πρόκληση θα είναι να συνεχιστούν οι εργασίες στους κόλπους του Συμβουλίου προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κατανόηση και να επιτευχθεί πρόοδος. Εφόσον λοιπόν εφαρμόσουμε τα όσα έχουμε συμφωνήσει, θα πρέπει παράλληλα να διευκρινίσουμε και να σιγουρευτούμε ότι η μετανάστευση θα παραμείνει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Χρειάζεται, ξέρετε, ένα σύστημα βιώσιμο για πιο δίκαιη κατανομή των βαρών και θα πρέπει να έχουμε υπόψη την ανάγκη μεταρρύθμισης της συνθήκης του Δουβλίνου. Επίσης θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να δώσουμε συνέχεια σε όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο της Βαλέτα για την μετανάστευση και να εμπλέξουμε και κάποιες τρίστες χώρες σε ό,τι αφορά δηλαδή τις αιτίες της μετανάστευσης και κάποια ενδεχόμενη καλύτερη συνεργασία. Έχουμε και ευκαιρίε μπροστά μα. Έχουμε για παράδειγμα την ενιαία αγορά, που θεωρούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει πραγματικά να αξιοποιήσουμε το πλήρε δυναμικό τη και να αναπτύξουμε και την ε, ψηφιακή αγορά. για να πετύχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τις οικονομίες, για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρίως βελτιώνοντας την πρωτογενή νομοθεσία η οποία βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση και διάφορα θέματα θα επεξεργαστούμε στο πλαίσιο αυτό την Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση κεφαλαίων. Τώρα, σε θέματα ασφάλειας. Και αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Και οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν φρίκη και έγιναν αισθητέ παντού στην Νίκαια, στο Περολίνο, στις Βρυξέλλες. Προφανώς προκαλούν ανησυχία και ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πάντα σε θέση, να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση για να ε, εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας και σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο προφανώς μεταβάλλεται διαρκώς θα εργαστούμε για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση περιφερειακών αλλά και παγκόσμιων ζητημάτων. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική διπλωματία αποτελεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου η Ένωση να εστιαστεί στις δράσεις αυτές και θα συνεργαστούμε και με την υπηρεσία εξωτερική δράση. Τώρα, για θέματα κοινωνική συμπεριλήψη, η Μάλτα είναι εξαιρετικά περήφανη για το ιστορικό ρεκόρ που κατέχει εδώ και μπορούμε προφανώς θεωρούμε να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας και με τα επιτεύγματα μα θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία άλλωστε και με τις ΜΚΙΟ και με άλλες οργανώσεις για να συνεχίσουν να προαγάγονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των ε, ευάλωτων ομάδων, αλλά και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, για να συνεχίσουν να έχουν ε, ίση πρόσβαση σε... στην αγορά. Τώρα, οι γειτονικέ χώρες της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί μια περαιτέρω προτεραιότητα. Μεταξύ άλλων, προτεραιότητα αποτελεί και ο κλάδος της ναυτελίας, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξη. Και τώρα να πω δύο λόγια για τα σχέδιά μα σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, αν επιτρέπετε. Οι προσπαθίε μας θα εστιαστούν γύρω από δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να συνεχίσουμε ένα νομοθετικό έργο το οποίο λαμβάνει η χώρα σε τεχνικό επίπεδο στην παρούσα φάση και κυρίως αναφέρομαι στι διατάξει ESI του κανονισμού Omnibus όπου ελπίζουμε να πετύχουμε καλή πρόοδο. Υπάρχουν όμω και άλλα νομοθετήματα τα οποία είναι συζήτηση και τα οποία είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε στην Προεδρία μα. Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο που έχει να κάνει με τον κανονισμό όμνιβα, θα συνεχίσουμε την πρόοδο που ξεκίνησε η Προεδρία τη Σλοβακία. Η Σλοβακική Προεδρία πριν από εμά. Θα συνεχίσουμε το τεχνικό έργο στα αρμόδια σώματα του, του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πρόοδο στον τομέα αυτό. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες θα επιφέρουν ε, περαιτέρω απλοποίηση του πλαισίου εφαρμογής για την κοινή διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και στο πλαίσιο αυτό η Μάλτα θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απλοποίηση και ο αντίκτυπος που μπορεί να σημαίνει για τους ε, δικαιούχους και για τα σώματα τα οποία εφαρμόζουν τα προγράμματα. Και ο σκοπός λοιπόν είναι να συνεχίσει η πρόοδο στον τομέα αυτό για να επιτευχθεί συμφωνία στο εσωτερικό του Συμβουλίου για τα βασικά προβλήματα που μπλοκάρουν. Ο δεύτερο στόχο είναι να γίνει μια πολιτική συζήτηση για το πώ τα αποτελέσματα τη πολιτική συνοχή μπορούν να καταστούν πιο ορατά από του πολίτε. Πώ μπορούμε να τα προβάλλουμε πιο πολλού πολίτε. Και στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά την πολιτική, τη μελλοντική πολιτική συνοχή μετά το 2020, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά στοιχεία. Καταρχάς θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών τόπου, έτσι ώστε να κατανοεί ο μεμονωμένος πολίτης το τι κάνει η Ένωση. Δεύτερος στόχος είναι η απλούστευση των πολιτικών για αυτού οι οποίοι εμπλέκονται και τρίτον να αναπτύξουμε μία στραμμένη προς το μέλλον πολιτική η οποία να εφεύρει καινοτόμες λύσεις για τις νέες προκλήσεις. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών πιο αποτελεσματικά και πιο έγκαιρα χρονικά. Λαμβάνοντας υπόψη το έλλειμμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το οποίο τώρα κάνουμε και την αντίληψη που έχει ο πολίτης για αυτό που κάνουμε, Σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να καλύψουμε την απόσταση ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες της με αυτό τρόπο. Η πολιτική συνοχής είναι κεντρικό συστατικό για την επίτευξη των στόχων μας. Και ναι να αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχής ε, αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο σαν επενδυτική πολιτική, είναι απαραίτητο η συζήτηση για την πολιτική αυτή, την πολιτική συνοχής, να έχει σαν βασικό στόχο τη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειες και την επίτευξη της κοινωνικής, της οικονομικής και της περιφερειακής συνοχής. Για την επιτυχή εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής θα πρέπει να αναγνωριστούν καταρχάς οι ε, μεμονωμένες ανάγκες κάθε περιοχής και να υπάρξει επίσης αρκετή ευελιξία στη στήριξη των πρωτοβουλειών οι οποίες καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος, μία μοναδική σύνταγη, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες όλων των κρατών μελών. Και εδώ ακριβώς είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία την οποία έχουμε και νομίζουμε ότι η πολιτική εδώ θα μπορούσε να γίνει ε, μέσω διευκόλυνσης για τα κράτη-μέλη και όχι να υπάρχει ένα πακέτο το οποίο να κάνει σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι πολύ μηχανιστικό σαν στόχος και δεν νομίζουμε ότι θα είναι ε, κάτι το οποίο θα πετύχει. Το one size fits all δεν ε, νομίζω θα μας καλύψει. Ούτε μας ούτε τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Η οποία θα πρέπει να καλύπτει, όπως είπα, τις τοπικές ανάγκες. Περαιτέρω, ε, και άλλες προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών για την κοινή διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Εδώ η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση ε, έχει απλοποίηση, έχει να κάνει πολλή δουλειά, όπως και οι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το streamlining και την αναθεώρηση του οικονομικού κανονισμού. Η απλοποίηση πρέπει να είναι το κέντρο αυτών των διαδικασιών και θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από μια μείωση του διοικητικού βάρους και από περισσότερη αναλογικότητα. Θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία να μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί από όλους τους εμπλεκομένους και τις ε, μικρομεσαίες μεταξύ αυτών. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε με προγράμματα τα οποία βαρύνονται ιδιαίτερα από, τις ε, δικητικές ε, ε, από τα δακητικά βάρη και τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο δίσκαμπτα. Θα πρέπει η πολιτική συνοχή να είναι σε θέση να απαντήσει ταχύτατα και αποτελεσματικότητα μέσω των στοχευμένων επενδύσεων εκεί όπου κυρίως χρειάζεται, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παραμείνει τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής και σημαντικό μέσο για τη στήριξη των κρατών μελών και της επιτυχίας του ευρωπαϊκού προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να λειτουργήσει σαν μια πολιτική στραμμένη στο μέλλον, η οποία να καλύψει τα προβλήματα της Ένωσης και να καταστήσει την Ένωση ικανή να βρει καινοτόμες λύσεις. Σήμερα λοιπόν μου ζητήθηκε ε, να ενημερώσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ε, προτεραιότητες μας, ε, τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Νομίζω ότι θα πρέπει τα δύο όργανα τα οποία εκπροσωπούμε, εμείς και εσείς, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπόλοιπους εταίρους, να πετύχουμε, έτσι ώστε να δουλέψουμε λοιπόν μαζί τους επόμενους μήνες και να πετύχουμε ακριβώς τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς ε, το συμφέρον ε, των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε. Thank you. Thank you very much, Mr. Χαίρομαι που η παρουσίασή σας ε, τροποτινά συνέχισε την συζήτηση την οποία είχαμε πριν, πριν έρθετε στην αίθουσα γιατί μιλούσαμε για την ε, ορατότητα της ε, πολιτικής συνοχής και για το πόσο σημαντικό είναι να εξηγήσουμε και να πληροφορούμε τους Ευρωπαίους πολίτες για αυτή την πολιτική. Και χαίρομαι που αναφέρατε αυτές τις προτεραιότητες. Τώρα θα, θα, ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κύριος Βανιστερόη. Καταρχήν, ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ε, ευκαιρία. Ε, ε, με εντυπωσιάζει το πρόγραμμά σας, θα πρέπει να πω. Γιατί δεν μας ενημερώσατε για, σε σχέση με, τα, με τους άλλους, το έργο των άλλων υπουργών και δεν έχετε καθόλου στοιχεία εν σχέση με το πώς προτίθεστε ε, συγκεκριμένα να εφαρμόσετε όλα αυτά. Θα ήθελα να έχουμε πιο συγκεκριμένες ε, πληροφορίες. Συμφωνώ μαζί σας ότι η ευκαιρία να τεθεί το ζήτημα της περιφερειακής ε, πολιτικής είναι σημαντική υπό την Σλοβακή Προεδρία έγιναν πολλά πράγματα ούτω ώστε να δημιουργηθεί μια νέα νοοτροπία, νέος τρόπο σκέψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στι πιο προηγμένες ε, περιφέρειες. Ε, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο άτυπων συνεδριάσεων που έγιναν ε, υπό την ε, Σλοβακική Προεδρία. Ε, και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνουν οι συζητήσεις ακριβώς σε υψηλότερο επίπεδο. Πώς θέλετε εσείς να το οργανώσετε αυτό και πώς θέλετε να ενσωματώσετε, να καλέσετε τα δικά μας, τα μέλη, τα μέλη της δικής μας Επιτροπής εδώ, ώστε να συμμετάσχουν σε, αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει μια τέτοια παράδοση ενεργού συμμετοχής ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που ελπίζουμε να συνεχίσει. Και θα ήθελα να φέρω κάποιε σκέψει σχέση με θέματα συνοχής. Πιστεύω ότι μετά το Brexit ε, και θεωρούμε ότι θα γίνει κάτι διάρκεια της δικής σας Προεδρίας θα πρέπει να υπάρξει μια, ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την ε, Προεδρία. Εάν ένα μέλος φύγει, θα πρέπει οι υπόλοιπε χώρες να αναπτύξουν μια ακόμα πιο, πιο ξεκάθαρο όραμα για τη συνοχή. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια ε, πιο ισορροπημένη εξέλιξη στην Ευρώπη. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα εθνικισμών και αυξανόμενου λαϊκισμού, κάτι τέτοιο είναι σημαντικό. Ε, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συνοχής που είναι εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση θα γίνει στη δική σας Προεδρία και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όσον αφορά την Ευρώπη 2020 για τις ε, περιφέρειες, για τις πόλεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάτι τέτοιο. Παρακαλώ να μας περιγράψετε πώς προτίθεστε να το οργανώσετε και πώς θέλετε να συμπεριλάβετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Και μια τελευταία παρατήρηση για την λεγόμενη ορατότητα. Συμφωνώ μαζί σας και όπως ε, είπε ο Πρόεδρος μας, ήδη το συζητήσαμε σήμερα. Ε, συγκεκριμένες ε, προτάσεις σε σχέση με το πώς μπορεί να συμπεριληφθεί στη διαδικασία Omnibus ούτω ώστε να υπάρξει αυξημένη ορατότητα για τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε στο επίπεδο των πόλεων, των περιφερειών, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας κλπ. Ε, πώς ε, θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα στους ε, αποδέκτες αυτών των κονδυλίων να ε, καταστήσουν ορατά τα αποτελέσματα, να μιλήσουν για τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό είναι θετικό, δεν πρόκειται για λαϊκισμό. Παρακαλώ να μας κάνετε μια συγκεκριμένη πρόταση επικοινωνία, επικοινωνίας, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Προεδρία της ε, Μάλτας να κάνει κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο επιπλέον δεν είναι, ε, δεν συνεπάγεται κανένα κόστος. Κυρία Κρέλ από τους Σοσιαλιστές, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ σε πολλά πόσα είπε ο Λάμπερτ και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και σας κύριε Μπόργκ ε, για το θέμα της ε, μετανάστευσης και του ασύλου και το ότι είναι μια δική σας προτεραιότητα. Και ε, θα συμπεριληφθεί στη δικασία Omnibus. Έχει ήδη προβλεφθεί για τον τομέα της πολιτικής συνοχής, η μεταναστευτική πολιτική. Και νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει με πλατιά πλειοψηφία. Είναι σημαντικά το όσο είπατε για την πολιτική συνοχή. Για την ορατότητα είπε κάποια πράγματα ο Λάμπερτ, αλλά και η πρόεδρό μα. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ μια παρατήρηση την εξή. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να ενισχυθεί η ορατότητα εδώ, από τις Βρυξέλλες. Γιατί η πολιτική εφαρμόζεται στις περιφέρειες αυτό το οποίο θεωρώ ότι χωλαίνει είναι η, ο ζήλος, η δέσμευση των χωρών να δηλώσουν ότι είναι διατεθειμένες κάθε ε, περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα εδώ που μας το αποδεικνύουν. Αλλά έχω την αίσθηση εδώ ότι βρισκόμαστε σε ένα mainstream της επανεθνικοποίησης και προβάλλεται το επιχείρημα ότι από τις Βρυξέλλες ε, δεν ε, έρχεται τίποτα θετικό. Και εμείς ε, θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι είναι το δικό μας μέλημα να το αποδείξουμε. Αλλά για να το πετύχουμε χρειάζεται και η βούληση, συγκεκριμένη βούληση, πολιτική βούληση των χωρών μελών. Έχετε μια ιδέα για το πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε μια τέτοια πρόταση στο πλαίσιο της συζήτησης για την πολιτική συνοχής. Και έχω και μια ερώτηση. Είπατε ότι χρειαζόμαστε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο όσον αφορά την πολιτική συνοχή και εδώ συμφωνώ πολύ μαζί σας. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακαμπτή η προσέγγιση εδώ. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό γιατί ε, στη νέα περίοδο έχουμε θεσπίσει τρεις ε, διαφορετικές κατηγορίες ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ε, περιφερειών. Και συμφωνήσαμε το προπολογισμό που είναι όλο και πιο ισχνό, να τον ε, επικεντρώσουμε στι προτεραιότητε. αλλά δώσαμε, ε, αφήσαμε την ευελιξία σε εκείνε τι περιφέρειες που το χρειάζονται επιτακτικά να, ούτως ώστε να εξοπλίσουν όλες αυτές τι προτεραιότητε. Πού θέλετε εσείς ε, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Ίσως θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε καλύτερα, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολύ καλά τι εννοείται ακριβώς με αυτό. Και μία τελική ερώτηση. Η Επιτροπή τέλη Ιουνίου θα διοργανώσει ένα φόρουμ συνοχής. Θα υπάρξει τότε μια πρώτη προσέγγιση εκ μέρου της Προεδρίας ή εκ μέρου του Συμβουλίου να κάνει μια παρουσίαση για, τις, ε, για την μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής γιατί διάβασα σε ένα κείμενο του Κυβερνοβουλίου ότι θα γίνει μια άτυπη συνάντηση για την πολιτική συνοχή. Ε, το χαρτί αυτό το πήραμε ε, τον Ιούλιο, το πήραμε από τη δική μας υπηρεσία. Δεν ξέρω, ε, έχετε εσείς υπόψη σας να προετοιμάσετε τις δικές σας θέσεις πριν από αυτή τη διοργάνωση του φόρουμ. Η κυρία Τόματσικ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εξ ονόματος ε, της Κροατίας ε, και του νησιού το οποίο προέρχομαι, θα ήθελα να πω το εξή. Ε, να σας πω ότι ξέρω το πόσο είναι να ζει κανείς σε νησί. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση στα ευρωπαϊκά νησιά. Τα peer-to-peer, τα RX, τέτοια εργαλεία, τα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την προώθηση καλών πρακτικών και για την ανταλλαγή απόψεων. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς θα φροντίσετε για τη βελτίωση της ζωής στα ευρωπαϊκά νησιά με την ψηφιοποίηση και την καινοτομία. Κύριε Φαμίλτεμπρουχ, από την Άρντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας για τη συζήτηση αυτή, γιατί όπως είπατε, πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής Είμαστε υπό πολύ, πολύ πίεση. Αναφέρθηκε το Brexit, ε, το οποίο θα επηρεάσει και την πολιτική συνοχή λόγω του οικονομικού mainstreaming σε ό,τι αφορά τι επενδύσει στην Ευρώπη και είπατε ότι στην Προεδρία σα θα γίνει μια πρώτη γενική συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ε, πώς ε, θα το αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό, πώς θα φροντίσετε, θα γίνει λίγο πολύ μια συζήτηση συγκεντρωτική τον Ιούνιο και δεδομένη και τη Υπουργική Συνάντηση 8 και 9 Ιουνίου. Ποια είναι τα βασικά σημεία για την μετανάστευση, για παράδειγμα. Είσαστε διατεθειμένο να συζητήσετε και άλλα θέματα αρισιμότητα ε, μετά το 2020 για να συνηθούν οι βασικέ προτεραιότητε. Ε, όπως ε, είναι η στέγαση με τα μέσα τα οποία θα διατύφονται στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάτι πολιτικό ευαίσθητο το οποίο ενδεχομένω να βάλετε στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα συμμετέχει, το είπαν και οι συνάδελφοι, γιατί αν θέλουμε να σημειωθεί επιτυχία θα πρέπει και τα τρία θεσμικά όργανα να ε, δείξουν πρωτοβουλία και να σημειώσουν επιτυχίες. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ομαζή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μπόργκ για την παρουσίασή του. Αναφερθήκατε και σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, αναφερθήκατε δηλαδή στο γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκείτε την Προεδρία σας, αλλά δώσατε και κάποιες επιμέρους πληροφορίες για την πολιτική συνοχή. Είναι αλήθεια ότι το πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως είπατε. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, το Brexit είναι ένα θέμα και η οικονομική κρίση επίσης. Για το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης και για το θέμα της οικονομικής αιτίας των μεταναστευτικών ροών. Να μου επιτρέψετε να θυμίσω ορισμένους αριθμούς έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε τη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας. Το 2100 θα υπάρχουν στη γη 13 δις πολίτες. Το 2100 ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια. Και ταυτόχρονα το 2100 η Αφρική θα έχει τετραπλασιάσει τον πληθυσμό της από ένα δις που είναι σήμερα σε 4,2 δις. Το 2100 επαναλαμβάνει ο μιλητής. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν την οποία έχουμε μπροστά μας. Και δεν είμαι καθόλου μα καθόλου βέβαιος ότι οι λύσεις τις οποίες επεξεργαζόμεθα σήμερα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και εμείς άλλωστε, είναι το θέμα της συνεκτικότητας των κοινοτικών πολιτικών. Διότι εμείς δεν βρίσκουμε κανένα, δεν θα πετύχουμε κανένα αποτέλεσμα αν εφαρμόζουμε από τη μία πολιτικές οι οποίες καταστρέφονται από άλλες πολιτικές και αναφέρομαι εδώ στις εμπορικές ε, πολιτικές που έχουμε. Ένα δεύτερο σημείο και σας ευχαριστώ το, γιατί το αναφέρατε και ε, το έχουμε ήδη συζητήσει, είναι η ναυτική θαλάσσια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο νησιωτικός της εν μέρη χαρακτήρας. Δεν το έχουμε πει με ικανή επάρκεια αλλά από όλου τι υπήρου του κόσμου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία είναι η πολύ διασπασμένη, αυτή που έχει τα περισσότερα ανοίγματα θαλάσσια και με ένα τεράστιο αριθμό νήσων. Αυτό είναι ένα φυσικά σημαντικό πλεονέκτημα για την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη, ε, αυτό το οποίο θα ονομάζαμε δηλαδή ε, η γαλάζια οικονομία. Και γι' αυτό περιμένουμε από την δική σας Προεδρία λοιπόν να εμείνει περισσότερο στην θαλάσσια λιμενική διάσταση και επίσης ε, ε, στο θέμα των αστικών περιοχών, των μεγάλων πόλεων και μητροπόλεων. Απαιτείται λοιπόν εδώ να υπάρξει μια ενιαία στρατηγική για τα μέσα τα οποία έχουμε και για τις νησιωτικές περιφέρειες. Έρχομαι τώρα στα της πολιτικής συνοχής. Πριν να έλθετε στη συνεδρίασή μας σήμερα, είχαμε, είχε προηγηθεί ε, μία συζήτηση για το ΕΦΣΥ. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, ε, διαβλέπουμε μία ανησυχία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Έχω την αίσθηση ότι όσο λιγότερο καλά πηγαίνει η Ευρώπη, τόσο περισσότερο έχει ανάγκη από τη συνοχή. Όσο εξασθενεί η Ευρώπη, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει από την αλληλεγγύη. Αναρωτιέμαι όμως αν στο εσωτερικό του Συμβουλίου οι περισσότερες χώρες συμμερίζονται την άποψη αυτή και ποιοι είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο εσωτερικό του Συμβουλίου έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς την συνοχή. Γιατί αλλιώς το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν βαδίζουμε πλέον προς μια ιστορική παλινοδία, μια ιστορική υπαναχώρηση. Και αναρωτιέμαι αν θα βιώσουμε εμείς σαν κοινοβουλευτική εντολή τα βήματα αυτά τα αρνητικά για την περιφερειακή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τον κύριο Υπουργό για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή μας ε, και για την παρουσίασή του έχετε θέσει δύο βασικούς στόχους ό,τι αφορά την, ε, πολιτική συνοχή. Γιατί ως τώρα στις προεδρίες δεν υπήρχε τόσο πολύ η αναφορά στην περιφερειακή πολιτική. Ήταν πιο πολύ μια υποσημείωση η περιφερειακή πολιτική στο Ταμείο Επενδύσεων. Χαίρομαι λοιπόν που το αναφέρετε αυτό επισταμένος. Ρωτήσεις έχουν να κάνω για τρία θέματα. Πρώτο θέμα. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Ένα από τα θέματα προτεραιότητά σα. η μετανάστευση. Υποστηρίζω φυσικά την ανάγκη εξέβρεση ευρωπαϊκών λύσεων για τι ανθρωπιστικέ χρήσει και για τι γενικότερε ανθρωπιστικέ χρήσει και τις κρίσεις μετανάστευση, Μια κλίδα κατανομή και άμυνα. Στην πολιτική συνοχή επιμείναμε ιδιαίτερα από την Επιτροπή μας να ανοίξουν τα ταμεία και να ταχθούμε πιο πολύ υπέρ ε, των έργων ένταξης ε, και ενσωμάτωση στα πλαίσια και του κανονισμού Omnibus που αναφέρεται. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον έχετε θέσει συγκεκριμένε ε, πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αυτές οι λύσεις και αυτά τα μέσα από τα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι ως τώρα υπήρχε δυνατότητα από τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα λειτουργικά τους προγράμματα σε ό,τι αφορά τον τομέα το μετανασ... της μετανάστευσης, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα ένθερμη η υποδοχή από πλευρά των κρατών μελών. Γι' αυτό θεωρώ ότι μία ενημέρωση μια προβολή θα ήταν απαραίτητη, όπως είπατε. Το δεύτερο θέμα που αφορά και αυτό την προβολή του ζητήματος. Στην ε, Επιτροπή έχουμε κάνει μια τέτοια έκθεση, μια γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά την προβολή αυτής της αρχής εταιρικής σχέσης στην πολιτική συνοχή. Μεγάλο επίτευγμα για τη συμπερίληψη των τοπικών και περιφερειακών φορέων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών. Πείτε μας, αυτή η πολιτική εταιρική σχέση, ε, αυτή η εταιρική σχέση σας βρίσκει σύμφωνο τον υποστηρίζετε για τις στρατηγικές επενδύσεις που αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο της ε, πολιτικής αυτής. Προβλέπετε από πλευράς του Συμβουλίου Πρωτοβουλίας. Τρίτη ερώτηση, σύντομα. Από τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας δεν βλέπω τίποτα για τον Brexit. Μήπως το διάβασα καλά. Η επίκληση του άρθρου 50 θα γίνει στην Προεδρία σας και θα έχει ασφαλώς επιπτώσεις ε, στην περιφερειακή πολιτική και τη συνολική πολιτική σας. Για πείτε μας δύο λόγια λοιπόν και για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, η κυρία Ντεμάτο. Κύριε Υπουργέ, όπως το μαρτυρούν και οι διάφορες τροπολογίες και σε επίπεδο επιτροπής και στην Ολομέλεια, το κίνημα των πέντε αστέρων εξ ήταν κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Ε, ελπίζω η νέα σας κυβέρνηση να προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν και γι' αυτό το ερώτημά μου. Σύμφωνα με το άρθρο 16, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει, ε, να θέσει προς επανεξέταση τα συγκεκριμένα άρθρα και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει το αίτημα αυτό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να συνοδεύεται από μια νομοθετική πρόταση. Οι συνθήκες ε, το επιτρέπουν να κάνετε μια τέτοια πρόταση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Έχω τρεις επιπλέον ομιλητές στον κατάλογό μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στους συναδέλφους και μετά θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όλοι γνωρίζουμε ότι τους επόμενους μήνες ε, έχουμε σημαντικά θέματα για την πολιτική συνοχή. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον της πολιτικής αυτής, ένα πράγμα μετράει είναι το θέμα της απλοποίησης. Ανάμεσα στις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν για την απλοποίηση, τίθεται το θέμα της διαφοροποίησης στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Από τη μία δηλαδή στα πλαίσια της εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι οι δυσκολίες ίδιες για τους καλούς και κακούς μαθητές και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με το ύψος των πιστώσεων και ανάλογα της φύσης, την φύση των διαχειριστών των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Συνεπώς λοιπόν, εσείς θα προωθήσετε αυτή τη διαφοροποίηση, τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Έχετε κάνει κάποιες σκέψεις γύρω από αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα. Με ικανοποίηση βλέπω τη σημασία την οποία δίδεται στις θαλάσσιες περιοχές και στην πολιτική της ναυτιλίας. Εγώ είμαι από παραθαλάσσια περιοχή και αυτό με ικανοποιεί καταρχάς θα ήθελα να μάθω αν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα υπάρξει μια πολιτική σημαντική δήλωση γύρω από αυτό και αν πράγματι έχετε κάποιες επιπλέον φιλοδοξίες για τα θέματα που άπτονται της ναυτιλίας και των θαλασσίων περιοχών. Κύριος Νοβακόφ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ε, βλέπω ότι αναλάβατε τόσο τεράστια ευθύνη και πραγματικά ε, ελπίζω να σταθείτε αντάξιος. Ε, αναφερθήκατε στο ζήτημα της απλούστευσης και θα ήθελα να υπάρξει μία τουλάχιστον συγκεκριμένη πρωτοβουλία ε, ή μια ομάδα εργασία που να ασχοληθεί με το θέμα της απλούστευσης και να αξιοποιηθεί η εμπειρία της Ολλανδικής ε, Προεδρίας. Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει ένα έγγραφο που να ε, ζητά μεγαλύτερη απλούστευση. Δεύτερον, ποια είναι η στάση σας έναντι της, ε, ε uh, της καινοτομίας. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μία έλλειψη πόρων για το Horizon. Πώς ε, θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα και ποια είναι η στάση σας έναντι της ε, καινοτομίας εν του ισχνού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. δεν θα ήθελα να συζητήσω άλλες προτεραιότητες πλην της πολιτικής συνοχής και είμαι ευτυχής που στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ε, υπογραμμίσατε την εφαρμογή των στόχων του 2020 γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε ένα ψήφισμα και αυτή τη στιγμή εκπονείται ένα δεύτερο σε σχέση με την επιτάχυνση της εφαρμογής της, της πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε το εξής. Ε, προτίθεστε να αναλάβετε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε ή έχετε κάποιες προτάσεις για να επιταχυνθεί η εφαρμογή και πώς ε, θέλετε να προτείνετε στις χώρες μέλη να ξεπεράσουν τα πρακτικά εμπόδια που υφίστανται στο πεδίο της εφαρμογής. Και ε, τη τελευταία ερώτηση θα υποβάλει ο κ. Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία για μας για να σας διαβιβάσουμε τις ανησυχίες μας. Ελπίζουμε να είναι μια καλή Προεδρία για όλους. Ε, έγινε κατά επανάληψη λόγος για την πολιτική της συνοχής ε, στις χώρες μέλη επιθυμούμε την απλούστευση και την ε, επιτάχυνση της διευκόλυνσης μιας καλύτερης πρόσβασης. Από την άλλη θέλουμε μια καλύτερη ορατότητα της πολιτικής συνοχής και δικαιολογημένα υπογραμμίστε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα τα οποία γίνονται και χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη αλλά αχνώνονται από τους πολίτες. Άρα λοιπόν σε αυτό φταίει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο γιατί δεν είμαστε ικανοί να περάσουμε το θετικό μήνυμα να περάσουμε μια θετική εικόνα της Ευρώπης που δράει υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Έγινε λόγος για τη μετανάστευση και θα ήθελα να πω το εξή από την πλευρά της δικής μου χώρας, της Ρουμανίας. Νομίζω ότι είμαστε θύματα μιας μεγάλης αδικίας γιατί δεν συμμετέχουμε στη ζώνη Σέγγεν παρόλο που τα σύνορα είναι ασφαλή. Υπάρχουν άλλες χώρες των οποίων τα σύνορα δεν είναι τόσο ασφαλή όσο τα δικά μας και είναι μέλη του Σέγγεν, της ζώνης Σέγγεν. Θα ήθελα λοιπόν να αποστείλετε ένα ηχηρό μήνυμα ούτως ώστε να εξαλειφθεί αυτή η διάκριση θα έπρεπε να μπούμε στη, στο χώρο Σέγγεν, τουλάχιστον όσον αφορά τον εναέριο χώρο. Όσον αφορά τη βαρύτητα του μεταναστευτικού φαινομένου, προσπαθούμε στην Ευρώπη να δημιουργήσουμε κέντρα υποδοχής για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα για την περίοδο του χειμώνα και του μεγάλου ψύχους. Δεν θα ήταν όμως πιο χρήσιμο να υπάρξει, να γίνει χρηματοδότηση στις χώρες ε, προέλευσης των ε, προσφύγων, ούτως ώστε να μετατοπιστεί η έμφαση όχι στις δαπάνες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αλλά στις δαπάνες που γίνονται υπέρ των προσφύγων στις χώρες προέλευσής τους. Ευχαριστώ πολύ. Και ο λόγος των Υπουργών για να ακούσουμε απαντήσει. απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με πάσα ειλικρίνεια πρέπει να ομολογήσω ότι δεν περίμενα τόσο πολλέ ερωτήσει και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο να σα απαντήσω. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλε ευκαιρίε ε, για να συνομιλήσουμε. Είμαι αρμόδιο ω υπουργό Θα είμαι μάλλον ε, υπεύθυνο για τι συνόδου τη Ολομέλεια. Ε, θα τι καλύψω, θα τι καλύπτω εγώ. Και γι' αυτό και προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συζητήσει κατά τη διάρκεια τη Ολομέλεια. Ε, πέραν τούτου είμαι υπεύθυνο και για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και γι' αυτό λοιπόν παρίσταμε εδώ σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι συναντήσει, τι επίσημε και τι ανεπίσημε, το μήνυμα που θα αποστείλουμε Ω Προεδρία είναι το εξή. Θα δύο υπουργικέ ε, συναντήσεις. Αυτό το έχετε παρατηρήσει και εσεί. Έχουμε το Σύμβουλιο Γενικών Υποθέσεων για τη Συνοχή τον Απρίλιο, στις 25 Απριλίου συγκεκριμένα, όπω και έχει οργανώσει η Σλοβακική Προεδρία. Σε αυτή την περίσταση, λοιπόν, θέλουμε να εγκρίνουμε συμπεράσματα από πλευρά του Συμβουλίου. και θα εργαστούμε, θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για τα ζητήματα αυτά. Η πολιτική θα πρέπει να είναι μέλλοντος τραφής. Και θα πρέπει προφανώς να υπάρχει καλύτερη προβολή και επικοινωνία των μηνυμάτων μας προς τους πολίτες. Θα γίνει και μια ανεπίσημη υπουργική συνάντηση το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο συναντήθηκα με την Πρόεδρο και την ενημέρωσα για την διεξαγωγή Υπουργική συναντήση πριν από το Φόρουμ Συνοχής, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Κοινοβουλίου. Και έτσι οι πρόεδρος και το Κοινοβούλιο θα έχουν την δυνατότητα να διαβιβάσουν και τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους ε, παρατηρήσεις μέσα του φόρουμ, το οποίο και δεσμεύεται να απευθυνθεί και σε εσά αλλά και στον Πρωθυπουργό μας που επίσης θα συμμετάσχει. Και ναι, λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. για να μην είναι σποραδική και, και κατακριματισμένη η διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, να υπάρχει ένας μύτος, ένας συνδετισμικός κρίκος. Δεδομένου των προκλήσεων λοιπόν που αντιμετωπίζουμε και είμαι πεπισμένος από τις δικές σας παρεμβάσεις ότι η πολιτική συνοχή είναι έτσι περαιτέρω πιο σημαντική για τέτοια ζητήματα, γιατί η πολιτική αυτή μπορεί να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, τα λαϊκιστικά, οι λαϊκιστικές εκκλήσεις απευθύνουν ακριβώς και βασίζονται σε τέτοια συναισθήματα. Γιατί οι υπομονωμένες ή οι μειονεκτούσες περιοχές συχνά έχουν την εντύπωση ότι είναι εγκαταλειμμένες από τους πολιτικούς. Η πολιτική εντυπωση οτι ειναι καταλημμενε απο τους πολιτικους η πολιτικη λοιπον αυτη θα πρέπει να οδηγήσει σε τέτοια έργα τα οποία θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη μείωση των διαφορών αυτών. Αναφερθήκαμε στο πακέτο Omnibus στην επικοινωνία σε σχέση με το πακέτο αυτό και θα γιορτάσουμε την επέτειο του ESF πάρα πολύ σημαντικό ταμείο και αυτό, το κοινωνικό ταμείο. Και στο μπλοκ 3 συζητάμε ήδη τέτοιες δυνατότητες. Στο τμήμα 3 ασχολούμεθα με τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Και εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω την εξής παρατήρηση ναι μεν ε, προεδρεύουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ξεχνάμε ότι και σαν κυβέρνηση της ε, Μάλτα και ε, γενικότερα σαν μια κυβέρνηση μια συγκεκριμένη χώρας, καλούμεθα να συνεργαστούμε με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει ε, σε συνεργασία λοιπόν με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουμε τα συμφέροντα όλων των χωρών της Ένωσης και στον τομέα του ασύλου και στον τομέα της μετανάστευσης. Το Νοέμβριο του 2015 είχαμε ήδη συναντηθεί στη Βαλέτα, είχαμε καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις σε σχέση με τα θέματα της Αφρικής και ξέρετε ότι η Αφρική είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί ε, την λεγόμενη οικονομική μετανάστευση κατά κύριο λόγο και είχαμε καταλήξει σε ορισμένες συμφωνίες για το τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας. Στην συνάντηση κορυφής λοιπόν στην Μάλτα στις 3 Φεβρουαρίου οι πρωθυπουργοί θα επανέλθουν στα θέματα που είχαν συζητηθεί και στην Πρατισλάβα έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα θέματα της μετανάστευσης και στον τομέα των σχέσεων με τις τρίτες χώρες, τις χώρες προέλευσης. Έτσι θα αποδείξουμε ότι είμαστε σοβαροί και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια μεταναστών θα μπορούν να ακολουθούν αυτόν τον τραγικό δρόμο, αυτή την τραγική οδό, αναζητώντας άσυλο ή ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σχετικά τώρα με τα θέματα της διαφάνειας και σχετικά με τα θέματα των ελέγχων και σε συμφωνία με σας προσπαθήσαμε να δούμε με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους να τα δαπανίσουν με καλύτερο τρόπο. Και αυτό ισχύει και για την χώρα μου και για τα νησιά. Εμείς είμαστε ένα μικρό νησί, είμαστε μια μικρή χώρα μέσα σε ένα μεγάλο αρχιπέλαγος. Γύρω από την Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και νομίζω ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις, οι περιφερειακές ανισότητες είναι κάτι το οποίο θα έλεγα συνδέεται με το μέλλον των νησιών και τα νησιά φύγονται διότι έχουν ε, θέματα μετακίνησης, κόστους μετακίνησης, υποδομών ακόμα και ηλεκτρονικών υποδομών που πολλές φορές είναι πολύ πιο ασθενείς από ό,τι στις υπηρετικές περιοχές. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη τον νησιωτικό χαρακτήρα και αυτό είναι κάτι το οποίο φύγει θα έλεγα σχεδόν το σύνολο των κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται και σε σχέση με την πολιτική 2020, την Ατζέντα 2020. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί προς την κατεύθυνση αυτή και σαν Συμβούλιο και σαν Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τις εξελίξεις και να δούμε ακριβώς τι έχουμε μπροστά μας, τι μας περιμένει εν πάση περιπτώσει έτσι ώστε αυτά τα οποία θα συμβούν στο μέλλον και οι πιθανές κρίσεις οι οποίες θα συμβούν στο μέλλον να μην μας προκαλέσουν αισθήματα έκπληξης. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις αυτές και θα πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να χαράξουμε ξεκάθαρες προοπτικές. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να λειτουργήσουμε με προληπτικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφύγουμε αρνητικές εξελίξεις. Και τέτοιου είδους συναντήσεις νομίζω θα βοηθήσουν και η επίσημη συνεδρίαση ε, του Συμβουλίου και η ανεπίσημη, τα φόρα τα οποία δημιουργούμε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάνουμε ε, την δυνατότητα την οποία μας παρέχουν οι συγκεκριμένες αυτές συναντήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι ανησυχίες μας και πώς μπορούμε τις ανησυχίες αυτές να τις καλύπτουμε. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις εμείς καταγράψαμε τα σχόλιά σας, είδαμε τις παρατηρήσεις σας και ακούσαμε προσεκτικά αυτά τα οποία μας είπατε και για το Brexit. Εμείς περιμένουμε την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας του Brexit, οπότε δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι υποθετικό. Πάντως δεν πάβει να είναι μια επιπλέον δυσκολία την οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Πάντως είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο θα έλεγα είναι ενωμένο ε, με μία φωνή. Συνειδητοποιούμε ότι η καιρή μπροστά μας είναι δύσκολη, αλλά είναι και μια ευκαιρία για μας να είμαστε πιο ενωμένοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί είναι μια ειδική κατάσταση και σύντομα θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια της ευρωπαϊκής προοπτικής. Ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο θα συνεδριάσει σύντομα στην ε, Μάλτα, όπως και η συνάντηση κορυφής της 3ης Φεβρουαρίου, θα λειτουργήσουν με χρήσιμο τρόπο για να μπορέσουμε να αποστείλουμε ε, τα σωστά μηνύματα. έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να πετύχουμε. Μιλάμε για τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία 60 χρόνια η Ήπειρός μας εν πολλής έχει ζήσει ε, μια εποχή ειρήνης και ανάπτυξη. Ε, και πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης αναπτύχθηκαν, προόδευσαν, βελτιώθηκαν οι συνθήκες ζωής των πολιτών και ναι, να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, έχουμε όμως και πολλά θετικά τα οποία έχουμε πετύχει και τα οποία πρέπει να τονώσουμε ακόμα περισσότερο. Εγώ είμαι αρκετά νέος ηλικιακά, όπως είπε άλλωστε ένα συνάδελφό σας, αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα διατηρήσουμε το ενιαίο νόμισμα, το πλεονέκτημα του να ανήκει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι κοινέ προσπάθειες τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την Ευρώπη την οποία θέλουμε να βιώσουμε στο μέλλον. Λοιπόν, ε, ε, πάντοτε θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου ε, μια χώρα μέλος ενδεχομένω θα θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που μου θέσατε. Ε, ο τομέας της ναυσιπλοείας ναι, ανεφέρθηκε. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό εδώ που μπορεί να αξιοποιηθεί και θα θέλαμε να δούμε πώς θα εγκριθεί η σχετική στρατηγική. Επίσης όσον αφορά την γαλάζια ανάπτυξη, και την πολιτική που έχει αναπτυχθεί στον τομέα αυτό. Πολλές φορές ε, παραλείπουμε να αναφέρουμε το δυναμικό των ωκεανών και των ε, θαλασσών μας. Ε, συνήθως αναφερόμαστε στους ωκεανούς και στις θάλασσες όταν συμβαίνει κάποια τραγωδία. Παρ' όλα αυτά, ο τομέας αυτός έχει ένα τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την καινοτομία και Επίσης ε, υπάρχουν σχετικές αναφορές όσον αφορά τα ταμεία ε, και υπάρχουν και πολλές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασία ε, και τόμες ευκαιρίες. Πρόκειται για ένα τομέα που μπορεί να παράσχει τέτοιες ευκαιρίες και είμαι σίγουρος ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν πιθανότητες και σε άλλους τομείς ούτως ώστε να συζητήσουμε και θα υπάρξει και η ευκαιρία να ξανασυστήσουμε όλα αυτά τα θέματα και πιο συγκεκριμένα τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας της ε, Μάλτα. Στο τομέα αυτό αναφέρθηκα ήδη στην καινοτομία και έχω την αίσθηση ότι ε, μπορώ να συμφωνήσω με το γεγονός ότι όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά επίσης και την ε, ανάγκη δημιουργίας περισσότερων θέσεων απασχόλησης, έχουμε ανάγκη μια πιο καινοτόμο Ευρώπη. Ε, και οι λοιπές ήπειροι θέτουν προκλήσεις και πολλοί Ευρωπαίοι προσελκύονται από άλλες υπήρους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παγκόσμια πρόκληση εδώ και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα οικονομικά μέσα ούτως ώστε να στηρίξουμε τα καλά προγράμματα ε, κυρίως όσον αφορά και την ε, στρατηγική 2020 και τη φάση βεβαίως εφαρμογής. Θα πρέπει εδώ να αναγνωρίσουμε ότι έχουν ε, εμφανιστεί νέες προκλήσεις όπως οι στρατηγικές που είναι αναγκαίο να εκπονηθούν πριν από τη φάση της εφαρμαγής. Επίσης, το ζήτημα της αρισιμότητας των διαφορών κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να εκπληρωθούν. Επίσης, ε, δεν έχουμε ε, σήμερα όλες τις ε, αναγκαίες πληροφορίες από τις χώρες μέλη σε σχέση με τα ποσοστά δέσμευσης κάθε χώρας. Ε, ξέρουμε κάποιους ε, αριθμούς και γνωρίζουμε ότι οι χώρες μέλη κάνουν ό,τι μπορούν. Και βεβαίως εάν δεν υπάρξει κάποια επιτάχυνση θα χάσουμε την κατάλληλη ευκαιρία. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ούτως ώστε να πετύχουμε αυτή την αναγκαία επιτάχυνση. Βεβαίως στο πλαίσιο της Προεδρίας υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Θα συνεχίσουμε βεβαίως να εστιάζουμε στις προτεραιότητες αυτές και προσπαθούμε να κατανοούμε ε, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις εφόσον υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης τέθηκε μια ερώτηση σε σχέση με, με, τους, ε, με την αναστολή των υφιστάμενων ε, κανονισμών. Εγώ νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε στη βάση των παρόντων κανονισμών. Ω Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουμε μια δυνατότητα να συνεργαστούμε και να κοιτάξουμε προς το μέλλον για να αυξήσουμε την ορατότητα συνεργαζόμενοι επίσης και με άλλα θεσμικά όργανα. Εγώ έχω την ευκαιρία να δράσω, είχα μάλλον την ευκαιρία στο παρελθόν ως δήμαρχος να αναλάβω δραστηριότητα στην Επιτροπή Περιφερειών και θα διοργανώσουμε μελλοντικά δημόσιους διαλόγους, ούτως ώστε σε διάφορες πόλεις και περιφέρειες να μπορούμε να εξηγήσουμε πώς ακριβώς συστάθηκαν τα διάφορα προγράμματα, ούτε ώστε οι πολίτες να μην θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι δεδομένο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε τη φάση του σχεδιασμού καθώς και την συμμετοχή των πολιτών. Και εάν εσείς ως Επιτροπή έχετε την αίσθηση ότι μπορείτε να συμβάλλετε εδώ, να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω θα μπορούσαμε από κοινού να ε, διοργανώσουμε τέτοιου πρωτοβουλίες. Ενδεχομένως υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις τις οποίες ε, παρέλειψα, αλλά θα είμαι παρόν στις Ολομέλειες ε, του Στρασβούργου και θα βρίσκομαι και εδώ στις ε, Βρυξέλλες και θα είμαι στη διάθεσή σας να συναντηθώ μαζί σας και σε ατομικό επίπεδο εφόσον το επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις. Να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή μας είναι ιδιαίτερος φιλόδοξη και εστιαζόμαστε στην πολιτική συνοχή. Εργαζόμαστε για μία σύγχρονη αλλά και μία μελλοντική πολιτική συνοχή. Καλωσορίζουμε την απλοποίηση εξετάζουμε με κρατικό πνεύμα τι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο θα συνεχίσουμε τη συζητήση για την εφαρμογή της πολιτική συνοχή με τον Γενικό, Γραμματε, τον Γενικό Διευθυντή της DG Regio. Θα είμαστε πολύ αξιόπιστος λοιπόν και σοβαρός εταίρους για όλες τις ε, συναντήσεις που διοργανώνεται και τις εκδηλώσεις που διοργανώνεται στα φόρουμ, στις πλατφόρμες και το καθεξής. Έχετε λοιπόν εδώ πέρα μεταξύ μας υποστηρικτές, υποστηρικτές σε ό,τι αφορά τα σχέδιά σας για την πολιτική συνοχή. Και εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής μας σας εύχομαι με κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Ελπίζουμε να μπορέσετε να διαμορφώσετε μία ιδιαίτερα ορατή πολιτική με τις κοινέ μας προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Και πέρα στις συνεδρίες, τα λέμε αύριο το πρωί στις 9.